Ja, Kolleginnen und Kollegen, ich möchte dann die Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι σήμερα το πρωί της εργασίας μας και θα ακούσουμε τους προσκεκλημένους υπουργούς και με την Προεδρία της Δανίας. Χθες ακριβώς υποδεχτήκαμε την ε, Επιτροπο, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και αλίες και Αγροτικής Ανάπτυξης και σήμερα θα έχουμε την Πία Ολσεντήρ προσκεκλημένη η οποία και θα λάβει το λόγο μάλλον ε, επειδή αδυνατή να παραστεί θα έχουμε τον αντικαταστάτη της δεν θα ήθελα να καθυστερήσω άλλο και έχει το λόγο ο εκπρόσωπος της Δανέζας Υπουργού για να μας εξηγήσει ακριβώς τι μπορούμε να περιμένουμε από την Δανική Προεδρία. Θα ακολουθήσει δε συζήτηση. Έχουμε 10-15 λεπτά για την παρουσίαση και μετά οι συνάδελφοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις και θα έχουμε δεύτερη σειρά ερωτήσεων. Έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της Προεδρίας μας σε θέματα υγείας. Συμμετείχα επίσημα στην συνάντηση στην Κοπενχάγη και ο πρόεδρος τότε τεμπούζε ήταν παρόν και θα ήθελα να σας πω ε, και υπόθηκε ότι θα βρείτε φίλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σίγουρα αναφυσβήτητα χάρηκα πάντως που το έμαθα ότι εδώ θα έχω φίλους και είμαι έτοιμη να ξεκινήσω μια συζήτηση για θέματα υγείας και είναι η ενδέκατη ημέρα μου σαν ε, Υπουργό Υγεία και θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσω στην όλη συζήτηση και ανάπτυξη σκληρό έργο στο Συμβούλιο μετά από πολλές προτάσεις νομοθετικές που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται ε, ε, λοιπόν η βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χωρίς τη βοήθειά σας δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε κοινά αποτελέσματα υπέρ των ε, πολιτών της Ευρώπης και σε θέματα υγείας η Ιδανική Προεδρία επιθυμεί να πετύχει αποτελέσματα. Έχουμε τρία θέματα κύρια τα οποία μας απασχολούν τρεις τομείς ε, όπου μαζί θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε για τα 500 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα καινοτομία. Smart have better life. Οι εξύπνοι έχουν καλύτερη ζωή. Και αυτές ε, οι φροντίδες ε, να μην είναι μόνο οικονομικής φύσεως, είναι από τους καταλήτες ε, για καινοτόμες προσπάθειες στην Ευρώπη. Στην υγεία λοιπόν ε, περισσότερες προσπάθειες για να ξεφύγουμε και από την οικονομική κρίση. Δημογραφικές αλλαγές είναι πολύ σημαντικές. Χρειάζονται προσπάθειες ποιοτικέ για να ωφεληθούν οι ασθενείς. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή θέση όσον αφορά την παγκόσμια σκηνή χάρη στις καινοτομίες και η Δανία επιθυμεί να αναλύσει καλύτερα πώς θα μπορέσουμε να έχουμε καινοτομίες στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασκήσει μια κριτική βέβαια την διαχείριση την οικονομική για αυτές τις φροντίδες και αυτό ισχύει και για την ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να βελτιωθούμε για να βοηθήσουμε τους ασθενείς και τους καταναλωτές μέσω καινοτομιών όπως είπαμε. Και οι καταναλωτές ε, θα πρέπει να συμμετάσχουν στην διαδικασία για την εφαρμογή αυτών των καινοτόμων ιδεών. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ε, φροντίδες ε, ακριβώς και να βοηθάμε τους ασθενείς. Ε, απαιτείται ένα πλαίσιο κατάλληλο για τις καινοτομίες αυτές. Στην άτυπη συνάντηση την Υπουργική του Απριλίου, το Smarts Have Better Life, αυτό θα είναι στην ημερήσια διάταξη τον Απρίλιο ακριβώς και επίσης ε, την Μάιο την ε, εβδομάδα που θα φέρετε αυτά τα θέματα στην Κοπενχάγη. Όλα αυτά αποτελούν την προτεραιότητα επίσης της ε, δανική προεδρία με τις χρόνιες ασθένειε. Είναι μια πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη γιατί... Ε, πάρα πολλοί πολίτες στην Ευρώπη ζουν περισσότερα χρόνια και με μια χρόνια όμως ασθένεια. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το προσέξουμε, να δούμε πώς θα έχει η πρόσβαση σε ορισμένα, σε ορισμένα, σε ορισμένα φάρμακα, παρασχάρη για την περίπτωση του διαβήτη θα πρέπει να δούμε ποιοτική προσφορά και όπως είπαμε στην ασθένεια αυτή θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην όλη διαχείριση βάση της πείρας που διαθέτουμε για το διαβήτη και να δούμε μέσω αυτών των φροντίδων πώς αντιμετωπίσουμε και άλλες ασθένειες. Όλα αυτά λοιπόν για τον ασθενή και στην στήριξη των ασθενών Όσοι υποφέρουν από χρόνιες ασθένειες θα πρέπει να μπορέσουν να ζουν ποιοτικά και να αντιμετωπίζουν αυτές τις χρόνιες ασθένειες και σίγουρα και ηλεκτρονικά μέσα όλα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να είναι αυτόνομοι αυτοί οι ασθενείς. Να μην έχουμε μόνο ελέγχους νοσοκομεία και ε, να είναι η δυνατότητα ο καθένας να αντιμετωπίζει από μόνος του την ασθένειά του και να προχωράει κατάλληλα. Και επίσης ε, η αντίσταση των ε, μικροβίων θα πρέπει να δούμε πώς θα την κατανικήσουμε και χρειάζεται μια συνεργασία και από τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο χρειάζεται μια συνεργασία ανάμεσα θεσμικά όργανα του ε, της Ευρωπαϊκή Ένωσης και χαίρομαι που η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα θεωρούν αυτά ότι έχουν προτεραιότητα. Θα πρέπει να συμμετάσχει το Κοινοβούλιο στην όλη συζήτηση όπως είπαμε και εμείς επιθυμούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία και με τις κτηνιατρικές μονάδες επίσης εκτός από, τις ιατρικές, από τα ιατρικά τμήματα για αυτή την ανθεκτικότητα των μικροβίων. Θα πρέπει αυτή να μειωθεί στην Ευρώπη και επίσης χρειάζεται να δούμε τι κατάλληλα αντιβιωτικά θα χρησιμοποιούμε και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ε, τα ισχυρότερα αντιβιωτικά μόνο όταν είναι απόλυτα απαραίτητα θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα την κατανάλωση ακριβώς αντιβιωτικών, διότι προκαλούν ε, αυτή την ε, αντοχή στα μικρόβια, και 14 και 15 Μαρτίου θα έχουμε μια συνάντηση στην Κοπενχάγη για την μάχη αυτή και θα συμμετάσχουν εμπειρογνώμονες όπως και υπάλληλοι από τον ιατρικό τομέα και από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για να μπορέσουμε να δώσουμε μια κατάλληλη απάντηση σε αυτό το πρόβλημα. Σε συνεργασία βέβαια με τον ε, αντίστοιχο Υπουργό Κατανάλωσης και θα θέλαμε να ζητήσουμε την, την πολιτική σας υποστήριξη για αυτή την τόσο σημαντική μάχη που δίνουμε για να καταπολεμήσουμε την ανθεκτικότητα των μικροβίων στα αντιβιωτικά. Και η Δανία θα πρέπει να προχωρήσει σε πολλές ε, πρωτοβουλίες της Επιτροπής. Επίσης ε, μέχρι το 2020 με τις προτάσεις της Επιτροπής για τις ε, φροντίδες στους ασθενείς και επίσης ε, η υγεία είναι και μια αξία αλλά είναι και ένα σημαντικός καταλήτης για την ανάπτυξη. Θα προσέξουμε ιδιαίτερα γιατί σε τέτοιες περίοδους κρίσης θα πρέπει να υπάρχει η πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές, υψηλές ποιοτικές φροντίδες και όλα αυτά θα είναι δυνατά χάρη στην υιοθέτηση καινοτομιών και σε κατάλληλες φροντίδες όπως είπαμε και με νέες μεθόδους αποτελεσματικότερες για να μπορέσουμε να προλάβουμε προβλήματα υγείας και να ενισχύσουμε την υγεία και απέναντι επίσης και σε απειλές διαμεθοριακές σε θέματα υγείας Επίσης το θέμα αυτό θα το εξετάσουμε και η υποπολωνική προεδρία έχει ήδη εξεταστεί και ο αρμόδιος επίτροπος προχώρησε σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το πρόγραμμα αυτό και για να δούμε πώς θα συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας και με προστιθέμενη αξία βέβαια ευρωπαϊκή. Με την πρότασή μας προσέχουμε ιδιαίτερα αυτόν τον καταλήτη της ανάπτυξης. Θα πρέπει να πούμε ότι η υγεία είναι μια αξία αυτή καθ' αυτή. Υπό την Προεδρία μας ελπίζουμε ότι θα προωθήσουμε τη συζήτηση στην επόμενη συνάντηση που θα διεξαχθεί και τον Ιούνιο στο Συμβούλο ΕΠΣΚΟ θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Περιμένουμε και τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, και το Συμβούλιο έχει ξεκινήσει αυτές τις συζητήσεις. Έχουμε μια λεπτομεριακή συζήτηση που έχει διεξαχθεί και θα υπάρξει σίγουρα ένας διάλογος με τον Κοινοβούλιο και με τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα έχουμε ίσως τη δυνατότητα να κλείσουμε σε πρώτη ανάγνωση μια πρώτη συμφωνία. Ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί μια ε, συνεργασία, να υπάρξει μια συνεργασία που θα βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη. Και επίσης για τις απειλές της διαμεθοριακές σε θέματα υγείας θα το εξετάσουμε και αυτό στην, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Θέλουμε όλα αυτά να προχωρήσουν, ιδιαίτερα πριν από το τέλος του εξαμήνου της Προεδρίας μας. Γνωρίζετε ότι επίσης οι μολυσματικές ασθένειες δεν σέβονται τα σύνορα, δεν σταματούν στα σύνορα. Γι' αυτό ακριβώς και με τη βοήθεια της Επιτροπής θα καταβάλουμε προσπάθειες, όλα αυτά προετοιμάζονται και θα πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε κατάλληλα τη μάχη μας ε, κατά μελλοντικών κρίσεων σε παρόμοια θέματα. Και με εσά θα θέλαμε μια καλύτερη ευρωπαϊκή διαχείριση απέναντι στις απειλές κατά της υγείας και δεν ε, έχουμε τοποθετεί ακόμα όσο αφορά την πρόταση της Επιτροπής Ευρωπαϊκής, αλλά θέλουμε πάντως να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή προστασία όσον αφορά αυτές τις απειλές της διαμεθοριακής και θα πρέπει να έχουμε μία πρόταση για να ξεκινήσουμε την εργασία μας κατάλληλα και εδώ ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία με τις υπηρεσίες σας. Και όσον αφορά τα φάρμακα υπάρχει επίσης στο τραπέζι μία πρόταση από τον Οκτώβριο από την Επιτροπή στα πλαίσια μιας ευρύτερης συνεργασίας. Θα εξεταστεί όμως ξεχωριστά δέκα μετατροπές όσον αφορά τους κανονισμούς σχετικά με την επαγρύπνηση σε θέματα ε, φαρμάκων και θα υπάρξουν και σημαντικές αλλαγές για να βελτιώσουμε την αντιμετώπιση σε θέματα ασφάλειας φαρμάκων και μετά από την πρόταση, από μια κατάλληλη πρόταση, ε, πρώτα απ' όλα θα, για να αποσυρθεί ένα φάρμακο από την αγορά θα πρέπει να υπάρξει μια βαθιά ανάλυση και εξέταση του θέματος. Αυτά λοιπόν. Θα ήθελα να σας πω ότι θα μπορούσαμε πολύ σύντομα να ξεκινήσουμε συζητήσεις για όλα αυτά με το Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό. Ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις μας για την επερρύπνηση σε θέματα φαρμάκων υπό την δική μας Προεδρία και ελπίζουμε από δανεική πλευρά ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντο είναι έτοιμη να συνεργαστεί με γοργού ρυθμού μαζί μα. Ήδη πριν από 10 χρόνια υιοθετήσαμε διάφορους νέους κανονισμούς και ελπίζουμε γρήγορα να γίνει κάτι παρόμοιο και κατά τη διάρκεια αυτής της Προεδρίας μας αυτό και σχετικά επίσης με την ενημέρωση για τους ασθενείς, για τις συνταγές και υπάρχουν ορισμένες αφιβολίες και αντιδράσεις και διάφορες χώρες ε, εξέφρασαν δισταγμούς και αφιβολίες ε, όσον αφορά το θέμα αυτό σχετικά ε, με ορισμένες απαγορεύσεις που τις θεωρούν σαν αποκλεισμό δυνατοτήτων. Εδώ λοιπόν θα σας πούμε ότι θα υποβάλουμε προτάσεις για κάτι το σχετικό καινούριο θα θέλαμε να συζητήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα μπορούσε ίσως το κοινοβούλιο σας να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση και επίσης ε, για την οδηγία διαφάνεια τιμών και το θέμα αυτό το εξετάζουμε. Πρόκειται για μια οδηγία που έχει σαν στόχο να ισχύσουν προϋποθέσεις ε, ίδιες ε, για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, από το 1989 δεν έχει αλλάξει η σχετική οδηγία και από τότε έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και χαιρόμαστε για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζουμε να την ε, εξετάσουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς αυτής. Επίσης θα δούμε και πάλι την ομοθεσία για τους όλους χειρισμούς. Ε, και η Δανική Προεδρία θεωρεί αυτές τη, δυνατότητα μελέτης δηλαδή των προτάσεων ότι είναι εφικτή γιατί ε, διαθέτουμε χρόνο και αυτό με το Smart Have Better Life ε, αυτό μας απασχολεί και έχουμε αποφασίσει να προσέξουμε ιδιαίτερα τρία θέματα τα οποία μας φαίνονται ιδιαίτερα σημαντικά και είναι ήδη στη μερίσια διάταξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκινάμε έτσι μετά από τι εργασίε τη προηγούμενη ε, Προεδρία και σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πάντως θα μπορούσαν να συνεργαστούν ε, με αμοιβαία εμπιστοσύνη για ε, καταλληλότερες συνθήκες αντιμετώπισης προβλημάτων μαζί με τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκτενή αυτή παρουσίαση. Πολλά μας ε, παρουσιάσατε ως προτεραιότητες και τώρα θα ξεκινήσει ο γύρος των ερωτήσεων γιατί πρέπει να σας πω ότι έχω 14 συναδέλφους ήδη στον κατάλογο των ομιλητών. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Πέτρη Λίζα από την ομάδα του ε, ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να θέσω το θέμα των φαρμακευτικών προϊόντων, το οποίο μας απασχόλησε και χτες στην Επιτροπή μας, ε, με το σκάνδαλο συγκεκριμένα με τα... τα εμφυτεύματα ε, στήθους. Υπήρξε ένα παράδειγμα στην Δανία που καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι μετά από κάποια χρόνια να μπορούμε να εντοπίζουμε ποιο ε, είναι υπεύθυνο για την εμφύτευση αυτών των επιζήμιων επιβλαβών προϊόντων και σε ό,τι αφορά σε θέματα διανομής για να αποφευχθούν για παράδειγμα παραποιήσεις. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι το αμερικανικό μοντέλο, δηλαδή η καταχώρηση κάθε ενός ξεχωριστού προϊόντος και η έγκριση κάθε ενός ξεχωριστού προϊόντος αποτελείται σωστή οδό. Θα πρέπει να το συζητήσουμε. Δεύτερον, μιλήσατε για το Health for Growth, υγεία για την ανάπτυξη. Νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί. Φυσικά η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Όταν λέτε όμως ότι η υγεία δεν αποτελεί ε, αυτού αξία, νομίζω ότι αυτό θα έβρισκε αντίθετους ε, τους εκλογείς μας. Σε πέντε χρόνια δεν θέλει κανείς να έχει οικονομική ανάπτυξη, θέλει να έχει την υγεία του. Άρα λοιπόν θα έπρεπε ίσως να σκεφτούμε και θέματα που αφορούν και τον τίτλο. Ε, κοιτάξτε, σημαντική και η ανάπτυξη, αλλά και η υγεία χωρίς ανάπτυξη επίσης σημαντική είναι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε τέτοια θέματα τα οποία άπτονται τη υγεία των πολιτών μα. Τέλο, για την ενημέρωση των πολιτών. Εδώ η... το... το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πέρσι μία πρόταση για ένα fact box, αν θέλετε, ένα κυβότιο με πληροφορίες για τα πιο σημαντικά φαρμακευτικά, βιο... Ε, φαρμακευτικά προϊόντα σε ό,τι αφορά την επίδρασή του, τις παρενεργίες του κτλ. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με την ε, αντιμικροβιακή αντοχή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς και πολλοί βουλευτές μάλιστα, που θεωρούν ότι εντάξει όταν ε, πάυσουν αν θέλετε τα προβλήματα, μπορώ να σταματήσω να παίρνω τα αντιβιωτικά μου. Αλλά αυτό ακριβώς είναι αυτό που ενισχύει και η οικοδομία, αν θέλετε, την αντακτικότητα, την αντοχή στα αντιβιωτικά. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνει κανείς αντιβιωτικά του ακριβώς το χρονικό διάστημα το οποίο έχει προδιαγράψει ο γιατρός. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα και θα θέλαμε να συζητηθεί και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα είναι το Μακέβαν για τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ. Ο Πίτερ Λίζε ανέφερε τις ε, φαρμακευτικές συσκευές στα θέματα των εμφυτευμάτων. Έγινε λοιπόν μια συζήτηση χτες στο Κοινοβούλιο. Ακούσαμε πολλά από τα προβλήματα του συστήματος κωδικοποίησης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καταχώρηση στη χώρα μου, όταν ε, τελικά έπρεπε να διαπιστώσουμε ποιες γυναίκες ε, φέρουν ποια εμφυτεύματα, πολύ απλά κάποιες κλινικές δεν μπόρεσαν να μας βοηθήσουν. Σε άλλες περιπτώσεις είχαν καταχωρηθεί όλα τα εμφυτεύματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε χθε ότι κοιτάει και εξετάζει το ενδεχόμενο γραμμικών ε, κωδικοποιήσεων. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι το θέμα των φαρμαγευτικών συσκευών, των εμφυτευμάτων, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ πιο σοβαρά. Εμφυτεύονται στο σώμα των ανθρώπων και πείτε μου τι πιστεύετε για ενδεχόμενη πρώτερη έγκριση σε τέτοια περίπτωση συσκευών. Κάτι άλλο που προέκυψε. Η σχετική Αμερικανική υπηρεσία είχε έρθει σε επαφή με την ε, Γαλλική υπηρεσία το 2000, αλλά πολύ, καλά, πολύ απλά δεν είχε ενημερωθεί κανείς. Άρα θεωρώ ότι θα ήταν πολύ καλύτερο να υπάρχει ένα κεντρικό σημείο ενημέρωσης και πληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ε, ε, ιατρικές συσκευές. Πέρσι λοιπόν ξεκίνησα μια πρωτοβουλία, όπως θα γνωρίζετε, για την υγεία και διάφορες από τις διτάξεις θα εφαρμοστούν σύντομα. Η Προεδρία θα εξετάσει πώς εφαρμόζονται οι διτάξεις για την ηλεκτρονική υγεία, για παράδειγμα στα κρατημέλη. Το ίδιο ισχύει και για την ίδρυση εθνικών σημείων επαφής. Θα καταγράψει λοιπόν ε, η Προεδρία κατά πόσο έχουν προχωρήσει αυτά που συμφωνήσαμε σε ό,τι αφορά την φαρμακοεπαγρύπνηση και τη σχετική νομοθεσία για την, φαρμακευτική, για την ε, ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων. Ήμουν εισηγήτρια και θυμόμαστε ότι υπάρχουν τρία μικρά σημεία στο νόμο αυτό τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν. Και ξέρω ότι προσπαθούμε να περάσουμε σε μια γρήγορη πρώτη ανάγνωση, γιατί αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό για την δημόσια υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίντα. Για τους φιλελεύθερους τώρα, η Κορίν Λεπάζ. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για τις παρατηρήσεις που κάνατε. Τρεις ε, παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Υπάρχει ένα αυξανόμενο πρόβλημα που είναι αυτό των μακροχρόνιων ε, à tous ε, ασθενειών. Πολλές έχουν σχέση και με το περιβάλλον. Το θέμα της ε, πρόληψης και η σχέση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ του περιβάλλοντος στο οποίο εργάζεται κανείς και την κατάστασή του είναι κάτι το οποίο λαμβάνετε υπόψη στις μελέτες που κάνετε. Επίσης, αυτό που ανέφερε η κυρία Μακιον, δηλαδή το θέμα των PIP φυτευμάτων στις πλαστικές στήθους. Είναι ενδεχομένως ένα πρόβλημα για την Γαλλία, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Δηλαδή ότι υπάρχουν ε, οι προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική, τα οποία δεν έχουν περάσει από τον κατάλληλο έλεγχο. Και εδώ είναι θέμα δικαιώματος των ε, ασθενών, των καταναλωτών και θέμα προστασίας. Μπορεί κανένας να στραφεί κατά των ατόμων τα οποία δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα και να βοηθηθεί από την δικαιοσύνη. Τρίτο πρόβλημα, η θεραπεία με τα αντιβιωτικά. Μιλήσατε προηγουμένως για το θέμα αυτό. Υπάρχει μεγάλη αντίσταση στα αντιβιωτικά, όλο και περισσότερο. Μιλήσατε για το ότι το θέμα αυτό έχει σχέση επίσης και για την κτηνοτροφία. Προληπτικά χρησιμοποιούνται Cela rejoint également la question euh, des OGM, mais je pense que c'est votre... στην Έχει αυτό το θέμα της ε, προληπτικής χρήσης αντιβιωτικών στην ε, κτηνιατρική. Και τελειώνοντας, θα συμφωνήσω με τον Πίτερ Όκεν. Σε περιόδους μεγάλων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων και κρίσεων όπως η σημερινή, η υγεία είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό. Σημαντικό από οικονομικής πλευράς βεβαίως, αλλά δεν θα πρέπει κανείς να βλέπει πάντα το κόστος όσον αφορά την συλλογική υγεία, αλλά θα πρέπει να δει και την οπτική γωνία της ε, ε κοινωνικής, για την κοινωνική διάσταση και την ανθρώπινη διάσταση. Σε τέτοιες περιόδους για την υγεία του κανείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και σε αυτές τις περιόδους δύσκολες είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Κορίν και τώρα ο Καλ Σλίτερ και μετά η Ελέν Αντωνέσκου. Σας ευχαριστώ. Σας έθεσα δύο ερωτήσεις, ε, κάποιες ερωτήσεις ήδη, αλλά είναι δύο που δεν έχω θέση ακόμα. Ξέρετε ότι είχαμε ένα ψήφισμα τον Οκτώβριο για την αντιμικροβιακή εντοχή και μία από τις αξιώσεις που τέθηκαν είναι να σταματήσει ολοκληρωτικά οποιαδήποτε προληπτική χρήση, μόνο για θεραπευτική χρήση να χρησιμοποιούνται στην εκτροφή. Και δεύτερη πρόταση, να αναθεωρηθούν και να ανασταλεί η χρήση ε, αντιβιωτικών με, μη, με οργανισμού. τροποποιημένους οργανισμούς. Συγκεκριμένο ερώτημα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν γίνει ήδη δύο διασκέψεις για τις τιμές ε, και τη χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά τα κίνητρα για την κοινοτομία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ιατρική κοινοτομία, γιατί το κόστος το πληρώνει το κοινό. Και επίση δεν είναι θέμα σχετική αξίας, δεν είναι θέμα σχετικό. Δεν μπορεί να διαλέξει κανεί ένα καινούργιο κινητό ή το φάρμακο του για τον καρκίνο. Δεν υπάρχει επιλογή. Υπάρχει αυτή η διάκριση λοιπόν μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Και τι γίνεται με την παραγωγή χωρίς ε, υποχρεώσεις ε, άδεια, το οποίο θα ευνοούσε τους φτωχούς και θα ανταποκρινόταν στις ανάγκες της υγείας. Υπολογίστηκε το κόστος είναι δύο τρίτα του τι ξοδεύουμε για τα φάρμακα που, προ, που συνταγογραφούνται σήμερα. Σας ευχαριστούμε, Καρλ Σλούτερ. Η κυρία Αντωνέσκου. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα αρχίζοντας να εκφράσω την ικανοποίησή μου διότι βλέπω ότι η Προεδρία σας προσδίδει προτεραιότητα στις χρόνιες ασθένειες. Ξέρουμε ότι η επενδύσει για την καλύτερη διαχείριση των χρονίων ασθενειών μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των ασθενών και να ελαφρύνει κάπω το βάρο μια τέτοια ασθένεια για τον ασθενή, για την οικογένειά του, αλλά και για τα συστήματα υγεία. δεδομένου ότι σήμερα βρισκόμαστε σε δύσκολη οικονομική περίοδο. Οι ασθενεί, λοιπόν μπορεί να είναι αν θέλετε πιο ενεργοί για μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Θα ήθελα συγκεκριμένα να σας ρωτήσω το εξής ποια είναι τα διάφορα βήματα που θα λάβετε όσον αφορά την ε, πρόορη ε, αναγνώριση μέσω εξετάσεων κάποιων τέτοιων ασθενειών και ποια είναι τα σχέδια τα οποία έχετε για να μπορέσετε να βελτιώσετε τις ε, τράπεζες δεδομένων για τις ασθένειες μεταδοτικές ή όχι. Διότι χρειαζόμαστε βελτίωση των γνώσεων των οποίων έχουμε για τις χρόνιες ασθένειες. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω τη σχέση που υπάρχει μεταξύ υγείας και περιβάλλοντος. Το ανέφερε και μία συνάδελφος προηγουμένως. Ήδη είπαμε πόσο μας απασχολεί το θέμα των επιπτώσεων του περιβάλλοντος στην υγεία και κυρίως το θέμα της επιρροής των χημικών ε, ουσιών στην υγεία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, σας χαιρετίζω. Χαίρομαι για την Δανέζικη Προεδρία και ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας θα μπορέσουμε να κάνουμε νέα προγράμματα υγείας που θα βελτιώσει τα προγράμματα υγείας για όλε τις χώρες. Χαίρομαι που υπάρχει αυτή η πρώτη Κομισιόν, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο στην πρόληψη. Παρά το γεγονός ότι αναφέρεται η BCT, νομίζω ότι θα πρέπει γενικότερα να μιλήσουμε και για την διατροφή. Και νομίζω ότι η βιομηχανία των ειδών διατροφής θα πρέπει να αρχίσει να συνεργάζεται. Επίσης, στις, ε, για τον διαβήτη τύπου Β, νομίζω ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε αν υπάρχει καλύτερη διατροφή. Επίσης, το θέμα του καπνίσματος ε, και επιβλαβής υγείας του καπνίσματος είναι κάτι πολύ συναντημό. Και λυπούμε διότι όλο και περισσότερο καθυστερεί την οδηγία για τα προϊόντα καπνού η Κομισιό. Ελπίζω και διάρκεια λοιπόν τη Δανέζικη Προεδρία, κάτι θα κάνετε. Ξέρω ότι θα συνεργαστείτε εκ του σύνεγγυ για το θέμα αυτό με την Κυπριακή Προεδρία. Θα ήθελα να σα ερωτήσω ποια προληπτικά νομίζετε ότι μπορούμε και πρέπει να λάβουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση την ε, πρόληψη για θέματα υγεία. Ευχαριστώ. Ο Κρίστοφερ Φιέλνερ, ο οποίο είναι εισηγητή για την ενημέρωση των ασθενών. Κρίστοφερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πολύ που έχουμε χρόνο να πιούμε και ένα καφέ. Θα ήθελα, καταρχάς, να καλωσορίσω την κυρία Υπουργό Χαίρομαι ιδιαίτερα που ήρθατε να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες σας εδώ πέρα, γιατί μιλήσατε ιδιαίτερα και για την αντιμικροβιακή αντοχή, το οποίο είναι θέμα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα από τα βασικότερα προβλήματα υγείας, για το οποίο συζητάμε υπερβολικά λίγο, αν θέλετε, γιατί αποτελεί μια κοινή πρόκληση με την οποία ερχόμαστε όλοι αντιμέτωποι. Ελπίζω να συνεχίσετε λοιπόν το θέμα αυτό, να το εξετάζεται, αλλά να ασχοληθείτε και με την, ε, το, την υπόθεση των καινούριων αντιβιωτικών. Δεν θα ήθελα να επανέλθω σε αυτά που είπε ο κύριος Σλίτερ, αλλά νομίζω ότι στον τομέα των αντιβιωτικών θα μπορούσε να αναπτυχθούν καινούργια αντιβιωτικά και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια καινοτομία. Θα ήθελα να επισέλθω επίσης στο θέμα της ενημέρωσης, της πληροφόρησης για τα φάρμακα. Εδώ και πολλά χρόνια γνωρίζουμε ότι στο Συμβούλιο επικρατεί μεγάλη σκεπτικότητα για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπήρξε και μια πρόταση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία εγκρίθηκε μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Αλλά αυτή η διστακτικότητα, αν θέλετε, του Συμβουλίου δεν πρόκειται να εξαφανιστεί αν μείνουμε με τα χέρια δεμένα. Άρα θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θέλουμε να προωθήσουμε το θέμα αυτό, γιατί θα πρέπει να προσεγγίσουμε με επικοδομητικό τρόπο την πρόταση αυτή. Δεν είναι δυνατόν να καθόμαστε και να κοιμόμαστε και να θεωρούμε ότι με μια παθητική στάση θα εξαφανιστούν τα προβλήματα. Ξέρω ότι υπάρχουν και θέματα συνταγματικά και στην Δανία και στη Σουηδία σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Αλλά νομίζω ότι ακριβώς τέτοιου είδους προβλήματα θα πρέπει να, προσ... να προτείνουμε επικοδομητικές ε, λύσεις και θεωρούμε ότι η Δανία είναι από τις κατεξοχήν χώρες που εργάζονται με επικοδομητικό τρόπο. Άρα λοιπόν αυτό θεωρούμε ότι μας δίνει ευκαιρίες. Ευκαιρίες τις οποίες θα πρέπει να δράξουμε για να συζητήσουμε τις κοινέ μας ε, προσεγγίσεις. Εμείς από πλευρά Κοινοβουλίου είπαμε ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε τις, προ... τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την φαρμακοεπαγρύπνηση, αλλά ελπίζουμε ότι στο Συμβούλιο δεν θα το βάλουμε το θέμα αυτό στο ράφι, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί και η Ιδανική Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Τελευταία ομιλήτρια στον πρώτο ερωτήσεων. Και μετά θα μας απαντήσει η κυρία Υπουργό. Ε, I... Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να καλωσορίσω την Υπουργό. Θα σας ρωτήσω μία ερώτηση που δεν έχει να κάνει με νομοθετικά ζητήματα αυτή, αλλά ουσιαστικά με την ψυχική υγεία. Είμαι Ιρλανδή βουλευτής και συμμετέχω στο σχετικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ψυχική υγεία. Το σύμφωνο λοιπόν αυτό αναγνωρίζει τη σημασία της ψυχικής υγείας και θέλει να καταλήξει σε συστάσεις για ενέργεια σε πέντε τομείς. η πέντε αυτή είναι η πρόληψη των αυτοκτονιών και των ε, καταθλίψεων, ψυχική υγεία και εκπαίδευση, ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας, για να αποφευχθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και το στίγμα τι θα κάνει λοιπόν η Δανική Προεδρία για να δώσει συνέχεια με συγκεκριμένες δράσεις στο σύμφωνο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν λοιπόν ο πρώτος γύρος ερωτήσεων, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα να περάσουμε στις απαντήσεις της Υπουργού. Έχετε το λόγο. Τσακ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πολύ καλές ερωτήσεις, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Τον κύριο Λίζε πρώτα απ' όλα. Σχετικά με τα αμφιτεύματα στήθους και το σκάνδαλο αυτό, αρκετοί έχουν ήδη θίξει το θέμα, σίγουρα Σίγουρα θεωρούμε ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε μία ιδιαίτερη πρόκληση να αντιμετωπίσουμε σχετικά με τα φυτεύματα στήθους και όλοι μας θα θέλαμε να πετύχουμε μια λύση αλλά περιμένουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σαν Προεδρία εμείς ε, νομίζουμε ακριβώς ότι προχωράει στην ακτίμησή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη απόφαση αναθεώρηση γιατί υπάρχει έντονη ανησυχία ανάμεσα στον ε, γυναικείο πληθυσμό. Και ε, θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής. Θεωρώ ότι η υγεία είναι μια αξία αυτή καθευτή για τον καθένα από μας και σε επίπεδο οικογένειας, κοινότητας, και επίσης συμπληρωματικές αξίες ε, στα πλαίσια του θεμάτων υγείας και οι καταναλωτές παρομοίων συστημάτων ε, θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες να προχωρήσουν ε, σε καινοτομίες με νέα φάρμακα και σχετικά με παρασκευάσματα. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται ο πολίτης και αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει τη διαφορά αλλά και περισσότερο το χρησιμοποιούμε αυτό. Η ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία θα μπορούσε να επωφεληθεί από αυτή τη γνώση των ε, αναγκών των ε, πολιτών. Και κυρία μου, προσπάθησα να απαντήσω ε, προηγουμένως στο σκάνδαλο αυτό με τα εμφυτεύματα στήθους και σχετικά με τους κωδικούς εντάξει δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ιδιαίτερο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα ισχύσει αυτή η ασφάλεια την οποία χρειαζόμαστε σχετικά με τα εφητεύματα και για την φαρμακοεπαγρύπνηση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας για το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, να εξεταστεί γοργά αυτό το θέμα και μάλιστα με επικοδομητικό τρόπο. Πάντως ε, είμαστε ανοιχτοί απέναντι στο Κοινοβούλιο, περιμένουμε ότι όλα αυτά θα Μα ωφελήσουν και μας και σας. Κυρία Λεπάζ, ναι, απάντησα σχετικά με τα εφητεύματα στήθου, αλλά σχετικά με την υγεία συμφωνώ απόλυτα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όλα αυτά είναι σημαντικότατα για, εμά μας όλους και για τους πιο νέου και τους περισσότερο ηλικιωμένου. Και μιλήσαμε για την ενεργό γύρανση σε μια συνάντηση στην Κοπενχάγη γιατί και στο τέλος της ζωής ακόμα ε, είναι καλό οι πολίτες να μην ασθενούν ε, να είναι ενεργοί και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό για είναι μια ζωή με ιδιαίτερη αξία είτε είναι κανείς 15 ετών είτε 95 ετών και σχετικά με την ε, φαρμακοαντίσταση των μικροβίων. Εδώ θέλαμε μία στήριξη και να μπορέσουν να απαγορευθούν για προφύλαξη τα αντιβιωτικά. Ε, προχωράμε στις εργασίες μας, έχουμε ελπίδες. Κύριε Σλούτερ, μόλις μίλησα για την φαρμακοαντίσταση των μικροβίων, και επαναλαμβάνουμε, επαναλαμβάνουμε θα προσπαθήσουμε να μην χορηγούνται αντιβιωτικά για λόγους προφύλαξης. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα θέματα αντιμετωπίζονται και θα συναντηθείτε σίγουρα με αρμόδιους και θα τους υποβάλλετε τα ερωτήματά σας συζητήκαμε με την κοινοτομία. Κάθε φορά που έχουμε ένα νέο προϊόν, όλοι μπορούν να υποφεληθούν και οι πλουσιότεροι και οι φτωχότεροι. Δεν μιλάμε μόνο για φαρμακευτικά κατασκευάσματα, αλλά ε, ήμουν ας πούμε στη Ντουμπάι, στην κτίρια συνάντηση για φάρμακα και για ρυθμίσεις σε θέματα υγείας και μιλήσαμε για μια ειδική μορφή τουαλέτας. Ε, πολύ καλή που είναι μια εξέλιξη για τη βιομηχανία με δημιουργία θέσεων στην Ευρώπη και ταυτόχρονα και η ασθενείς θα μπορούσαν να υποφεληθούν. Άρα λοιπόν όλο αυτός ο συνδυασμός ε, ανάμεσα στην ανάπτυξη, στα νέα μέτρα, στα νέα προϊόντα είναι... μπορούμε να μιλήσουμε και για προστιθέμενη αξία. Και μια απάντηση τώρα για την κυρία Αντωνέσκου για τις χρόνιες ασθένειες συμφωνούμε. Πρόκειται για μια απόλυτη προτεραιότητα της Δανικής Προεδρίας θα πρέπει να διδαχθούμε ο ένας από τον άλλο με καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών γιατί να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις όλων μας για όλους και να προωθήσουμε το θέμα αυτό υπό Δανική Προεδρία. κυρία Γουίλμοτ, λυπάμαι που Κατακριούργησα το όνομά σας, λέει ο Μιλήτρια. Εδώ σχετικά με την υγεία μίλησα για αυτό το θέμα ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό για την Δανική Προεδρία και θα πρέπει να δούμε την πείρα που διαθέτουμε όσον αφορά θέματα διατροφής, ε, αθλημάτων, υνοπνεύματος, ε, ε, καπνού. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την υγεία. Όλα αυτά είναι και για τον διαβήτη Β, αλλά και για μια ολόκληρη σειρά άλλων ασθενειών. Γιατί πώς αν φερόμαστε στο σώμα μας, όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Εντάξει. Είμαι και υπουργό τη πρόληψη, εκτό από υπουργό υγεία, γιατί είναι κάτι το πολύ σημαντικό η πρόληψη στη Δανία και θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε, α πούμε, τον καπνό, το κάπνισμα, που είναι και η πρώτη αιτία θανάτων. Αλλά ελπίζουμε κάτι μπορούμε να κάνουμε και να το προχωρήσει αυτό βέβαια και υπό την Κυπριακή Προεδρία. Κρίστοφ Χέλνεν. Ε, χαίρομαι που χαίρεστε για την προσοχή που αποδίδουμε στην ε, φαρμακοαντίσταση των μικροβίων ε, και ελπίζουμε να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό και θα πρέπει όμως να λύσουμε το πρόβλημα που έχει να κάνει με την προληπτική χρήση αντιβιωτικών και Επίσης ε, για την ενημέρωση για τα φάρμακα υπάρχει ένας κάποιος σκεπτικισμός ε, στις τάξεις του Συμβουλίου και η δική σας ερώτηση είναι μια πρόκληση για τις κυβερνήσεις σας. Θα δούμε τι μπορούμε να έχουμε κάτι το θετικό σαν απάντηση. Πάντως είναι στα πλαίσια των όλων προβλημάτων. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, αλλά σας ευχαριστώ που λέτε ότι έχουμε επικοδομητική αντιμετώπιση εμείς στη Δανία και ότι θα προσπαθήσουμε σίγουρα να βρούμε μια λύση αυτά. Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Λυπάμαι, λυπάμαι κάτι, κάποιον λησμόνισα. Ναι, έχω πολλά χαρτιά μπροστά μου, πολλά φύλλα. Η κυρία Σέλντερτς. σχετικά με την διανοητική υγεία και την έκθεση του 2008. Όπως και άλλες προεδρίες, εμείς ε, επιλέγουμε προτεραιότητες. Μίλησα για τις τρεις μεγάλες προτεραιότητες. Αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε διάφορες μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις στον τομέα της υγείας και ταυτόχρονα στην εργασία μας ελπίζουμε να συνεργαστούμε με την προηγούμενη και με την επόμενη Προεδρία. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι θα πρέπει να θεωρούνται οι προτεραιότητές μας κάτι που αθρίζονται στις υπόλοιπες και όχι που απομακρύνονται, όπως είπε και η κυρία Σέλτερς. Αυτά τα προβλήματα τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Άκουσα την παρέμβασή σας και σημείωσα την απόψή σας. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ και να περάσουμε λοιπόν στο δεύτερο κύριο ερωτήσεων. Να ξεκινήσουμε με τον συνάδελφο Μύρος Λαφνικολάτσιτς που είναι ειδικό σε θέματα πολιτικής για την υγεία και μετά την κυρία Κάνμπαχ. Ναι, σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου, δεν είμαι σίγουρος γιατί οι συνάδελφοι με λένε Μικολάζε και συνάδελφοι από την γερμανόφωνο τομέα. Το όνομά μου είναι με S και K στο τέλος. Σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ που ήρθατε στην Επιτροπή μας, το εκτιμούμε ιδιαίτερα και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι σας βλέπουμε στο Υπουργείο αυτό. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι ακούσαμε το πολύ επικοδομητικό σας πρόγραμμα. Επιτρέψτε μου τώρα να θίξω κάποια ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν και να τα αναλύσουμε κάπως. Χτες συζητήσαμε το θέμα τον, του σκανδάλου των ε, εμφυτευμάτων σε πλαστικές τύθου. Μία γυναίκα η οποία επιθυμεί πλαστική στήθους και εμφυτεύματα έχει την ελευθερία να κάνει την επιλογή αυτή. Πολλές γυναίκες όμως από αυτές δεν συνειδητοποιούν ότι ενέχεται και ένας κίνδυνος. Το σύστημα λοιπόν θα έπρεπε να τις προειδοποιεί. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω και την Προεδρία σας να βελτιώσει την κατάσταση στον τομέα αυτό. Οι γυναίκες αυτές με δυσκολία θα μπορέσουν στο μέλλον ενδεχομένως να υποστούν διάγνωση για καρκίνο του στήθους, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολη η διάγνωση αυτή με το εμφύτευμα. Αυτά όλα είναι πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να έχει η κάθε γυναίκα στη διάθεσή της πρώτη αποφασίσει να προχωρήσει με την επέμβαση. Ασφαλώς αφενός αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα το οποίο και επιθυμεί να λύσει. Αφετέρου όμως τελικά συγκαταλέγεται σε μια ομάδα γυναικών οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα διάγνωσης ενδεχομένως στο μέλλον σε ό,τι αφορά καρκίνο του στήθους. Άρα θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η βασική προτεραιότητα είναι η υγεία. Κάτι άλλο, η ανείχνευσιμότητα. Αναφέρθηκε ένας γραμμικός κώδικας από την Λίντα Μακέβαντς. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να είναι δυνατή η ανείχνευση των προϊόντων αυτών για να εντοπίζεται κάθε συγκεκριμένο προϊόν. Συχνά στην Επιτροπή μας αλλά και στο σύνολο του Κοινοβουλίου συζητιέται το θέμα της σχετικής οδηγίας και κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα να εμπορευματοποιηθεί εν μέρη το ανθρώπινο σώμα. Νομίζω ότι και εσείς συζητάτε το θέμα αυτό και αν ακολουθήσουμε τις αρχές οι οποίες ίσχυαν ως τώρα, να μην εμπορευματοποιείται λοιπόν κανένα τμήμα του ανθρώπινου σώματος, αλλά παράλληλα να υπάρχει η δυνατότητα δωρεάς οργάνων, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση. Αυτή η αρχή λοιπόν θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσει, να εξακολουθήσει. Και θα ήθελα να καλωσορίσω την προτεραιότητα που θέτει η Ευρωπαϊκή η Ιδανική Προεδρία στις χρόνιες ασθένειες. Σημαντικός είναι και ο διαβήτης το θέμα αυτό, στο πλαίσιο αυτό. Να σας υπενθυμίσω ότι και εγώ έχω προβεί σε μια σχετική ανάλυση και στα 27-28 σύντομα κράτη-μέλη με την Κροατία πρέπει να διαπιστώσουμε ότι είναι πολύ διαφορετικές οι εθνικές νομοθεσίες σε ό,τι αφορά και την προστασία των μη καπνιστών. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν περαιτέρω και την έρευνα για τον αντίκτυπο του καπνού στην ανθρώπινη υγεία. Γιατί όλο και πιο πολλά άτομα ξεκινούν σε νεαρή το κάπνισμα, ιδιαίτερα γυναίκες σε κάποιε περιπτώσει μέχρι και 11 χρονών κοριτσάκια ξεκινούν το καπνίσμα, χωρίς να συνειδητοποιούν ποιο είναι ο αντικτύπο στην υγεία τους. Αν θα μπορούσατε λοιπόν να καλέσετε τα κρατημέλη να αναθεωρήσουν τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των μη καπνιστών. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος Θα τα καταφέρω καλύτερα την επόμενη εβδομάδα, είναι και πρώτη εβδομάδα, καταλαβαίνετε. Η κυρία Κάρμιν Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργέ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που, όπως και οι συνάδελφοί σας χτες, θέτετε την ε, καταπολέμηση της αντιμικροβιακής αντοχής και που στο πλαίσιο αυτό προτείνεται μια συνολική προσέγγιση. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ, να συνδυάσουμε και τον τομέα τη ιατρικής και της κτηνιατρικής. Να δείξω κάτι άλλο. Ο επίτροπο Ντάλι για... Στην... στον αγώνα του για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μη καπνιστών τον υποστηρίζουμε. Και να θέσω επίσης το θέμα της ανασωπήσης. φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, ε, τα εμβόλια έχουν καταστεί θύματα της ίδιας τους της επιτυχίας, γιατί αρρώστιες που θεωρούσαμε ότι θα είχαν εξαφανιστεί ε, μέχρι το 2020, τελικά βλέπουμε ότι δεν έχουν εξαφανιστεί και αυτό εν μέρει οφείλεται στις ε, λανθασμένες πληροφορίες που λαμβάνουμε από το διαδίκτυο και στην ελληπή ενημέρωση, αρρώστησε όπως η Λαρά για παράδειγμα. Η Ουγγρική Προεδρία τάχθηκε και εξέτασε αντίτρα το θέμα αυτό. Διοργάνωσε και μια διάσκεψη στην Βουδαπέστη. Στην τελευταία Προεδρία, ωστόσο, χαλάρωσε κάπως η επικέντρωση στο θέμα αυτό θα επικεντρωθείτε εσείς στο θέμα αυτό του εμβολιασμού των παιδιών για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν στα πλαίσια της Δανικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η Μαργρέτα Άουκ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και χαίρομαι επίσης που αντιμετωπίζει δύο διαφορετικά θέματα, αλλά σίγουρα θα σε στηρίξουμε. Και ελπίζω να σε στηρίξουν και οι όλοι οι υπόλοιποι. Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής. Κάτι που αφορά θέματα ακριβώς υγείας. για την κατανάλωση φαρμάκων. Πολλά φάρμακα καταλήγουν ε, στο περιβάλλον. Και αυτό επηρεάζει και τη δημοσία υγεία. Έχετε εξετάσει με ποιο τρόπο θα μπορούσε κανείς να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Την διάχυση των φαρμάκων στο περιβάλλον πώς να το πω τώρα, δηλαδή πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί το πρόβλημα αυτό με περισσότερο λογικό τρόπο από ό,τι μέχρι σήμερα. Γιατί κάτι που πάει στο περιβάλλον θεωρούσαν μέχρι τώρα ότι εντάξει πάει, έφυγε, χάθηκε. Δεν είναι όμως αυτό. Αλλά λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστούμε Άουκεν, Σοφία Μάτσεκ και μετά Hvala lepa, gospod predsednik, in lep pozdrav gospe ministrici. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον, την Υπουργό. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσίασή σας αυτή. Μίλησατε και για οικονομική ανάπτυξη. Πρώτα όμως ε, θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει καλή υγεία και πολλός κόσμος ασθενεί και λόγω της οικονομικής κρίσεως επειδή έχασε τη θέση του, δεν εργάζεται πια. Λοιπόν, πώς ε, θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε μια καλύτερη διαχείριση στο σύστημα υγείας. Υπάρχουν ιδιαίτερα περιθώρια για τη βελτίωση του συστήματος υγείας και μετά για να είναι κάτι τέτοιο αποτελεσματικό δεν θα πρέπει να έχει να κάνει μόνο με τον ασθενή και να είναι εις βάρος του ασθενή. Θα πρέπει να είναι μια καλύτερη εσωτερική διαχείριση, οργάνωση του συστήματος υγείας. Η υγεία. Η υγεία είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο. Γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να χαρακτηρίζεται από μια σφαιρική προσέγγιση απέναντι στον ασθενή. Σε λίγο οι ασθενείς θα μπορούν να, πηγαίνουν ελεύθερα από το ένα κράτος στο άλλο και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια μέτρα θα λάβετε για ένα συντονισμό και για μια ανταλλαγή στοιχείων πληροφοριών στο σύνολο της Ευρώπης, παραδείγματο χάρη για τις χρόνιες ασθένειες. Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Θα προσπαθήσετε να ελαφρύνετε το οικονομικό βάρος, έτσι, στο σύστημα υγείας. Και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ παραδείγματο χάρη στην ανάγκη συνταγογράφησης στην υπερβολική είτε για τις α, ε, μακρές ουρές αναμονής ε, εξετάσεων σε εργαστήρια. Και ακόμα, τι θα μπορούσε κανείς να κάνει όσον αφορά την πολιτική, την πολιτική υγεία, την οικολογική κλπ. σε τέτοια στιγμή κρίσης οικονομικής προβλέπεται συγκεκριμένα μέτρα και το πώς θα προχωρήσει κανείς στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά ας πούμε τη χρήση σιλικόνης που έχει καταντήσει να είναι μόδα πια και θα ήθελα να σε ευχηθώ καλή και αποτελεσματική εργασία και ελπίζω στα συμπεράσματά σας και συμπεράσματα του Συμβουλίου Υγείας να μπορέσετε να βελτιώσετε την κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να τηρήσουμε όμως πλέον το όριο των δύο λεπτών, προκειμένου όλοι όσοι είναι στο κατάλογο των αμελητών να έχουν την ευκαιρία να θέσουν τις ερωτήσεις τους και προκειμένου να έχει χρόνο και η Υπουργό να απαντήσει καταλήλως, γιατί ε, έχουμε και ένα χρονοδιάγραμμα. Dan Jürgensen. Και μετά η Άνια Βάισκερπερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Χαιρόμαστε που είστε εδώ σήμερα. Έχω δύο ερωτήσεις να σας κάνω. Η πρώτη έχει σχέση με ένα θέμα που αφορά και την πολιτική περιβάλλοντος και την πολιτική υγείας. Ξέρω ότι ασχολείσαι με θέματα υγείας, αλλά ασχολήθηκε με τα προβλήματα και ελπίζω ότι θα μπορέσει να μας απαντήσεις. Πρόκειται για το κοκτέιλ των χημικών προϊόντων. Υπάρχει η σχετική κοινοτική οδηγία και περνούμε από τις επικίνδυνες ουσίες τις λιγότερο επικίνδυνες, αλλά το, το κοκτέιλ αυτό που δημιουργεί η χρήση διαφόρων ουσιών που καταλήγουν σε πιο επικίνδυνο προϊόν δεν είναι ένα θέμα που έχουμε μελετήσει ακόμη. Προβλέπει η Δανική Προεδρία να μελετήσει το θέμα αυτό του σορευτικού αποτελέσματος χρήσης διαφόρων, ίσως όχι πολύ επικίνδυνων ουσιών, αλλά που συσσωρευόμενες μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνες. Σε μία άλλη επιτροπή μιλήσαμε για την πρόληψη του διαβήτη. Το ανέφερες, μπορείς όμως να μας πεις συγκεκριμένα τι μπορεί να γίνει για αυτό το θέμα. Δεδομένου ότι πάρα πολλοί πολίτες πιστεύουν ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε την παχυσαρκία, να έχουμε μια καλύτερη διατροφή, αλλά και ο διαβήτης είναι πάρα πολύ Ευχαριστώ. Η, κυρία Βάισπερκερ και μετά η Ροζα Σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Σας ευχαριστώ που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Χαιρόμαστε και εμείς ιδιαίτερα και προσβλέπουμε στη συνεργασία με την Προεδρία της, ε, του Συμβουλίου, επειδή έχω ιδιαίτερα στην εντύπωση ότι πρόκειται να διαδραματίσετε πολύ επικοδομητικό ρόλο και να προχωρήσετε με πολλά θέματα. Ένα θέμα που με απασχολεί ιδιαίτερα είναι και ένα θέμα το οποίο ανέφερε ήδη ο συνάδελφος Φιέλνερ αφορά την ενημέρωση, την πληροφόρηση των πολιτών. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν στο Συμβούλιο καταφέρνατε να ασχοληθείτε εντατικά με το θέμα αυτό και να βρείτε και κάποιες λύσεις. Θέλουμε να διαχωρίσουμε ένα σημείο, κάποια σημεία τα οποία ήταν πολύ σημαντικά για το Συμβούλιο από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θέλουμε να προωθήσουμε θέματα πληροφόρησης των ε, ασθενών. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να λαμβάνουν οι ασθενείς τι απαραίτητε πληροφορίε και θα ήθελα να σας δώσω κάποια επιπλέον επιχειρήματα. Πάνω από 50% των πληροφοριών τις οποίες βρίσκει κανείς στο διαδίκτυο σήμερα είναι εσφαλμένες και πολλοί ασθενείς χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να έχουμε ελεγμένες πληροφορίες στις οποίες να μπορεί να εμπιστεύεται και ο ασθενείς. Ε, σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν και κάποιες νομικές αμφιβολίες. Για παράδειγμα, στη Γερμανία έχουν παρουσιαστεί κάποια τέτοια ζητήματα. Θα μπορούσα και εγώ λοιπόν να φανταστώ ενδεχομένη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται για την έγκριση ενός προϊόντος. Ίσως αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μία μορφή συμβιβασμού. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα και τώρα η κυρία Άσο Βέσλοντ και μετά η Σοφία Κονή. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την κυρία Υπουργό. Εδώ μπροστά είμαι. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να, συναντήσω με, να συμφωνήσω με τους συναδέλφους σε ό,τι αφορά την αντιμικροβιακή αντοχή. Ελπίζω να προχωρήσει το θέμα αυτό η Δανική Προεδρία και σε ό,τι αφορά την διάσκεψη η οποία προγραμματίζεται. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αν ακολουθήσουμε την κλασική μέθοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ απλά διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα δεν προχωράνε επαρκώς ή ότι προχωρούν, αν θέλετε, στην ε, ανθρώπινη ιατρική, όχι όμως στην ηχθρήνη ιατρική. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε πώς θέλουμε να πετύχουμε τη μείωση της χρήσης των αντιβιωτικών. Πολλά θέματα όμως θα πρέπει να αποφασιστούν και σε επίπεδο κρατών μελών και όχι σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε έναν άλλο τομέα λοιπόν, στον τομέα αυτό έχετε δηλώσει ότι είναι προτεραιότητά σας εκεί η Προεδρία. Ελπίζω λοιπόν να το ακολουθήσετε αυτό προκειμένου να δραστηριοποιηθούν πολύ πιο έντονα οι Υπουργοί υγεία γιατί μιλάμε για χημικές ουσίες που αφορούν, για παράδειγμα, και τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως τα παιδιά. Ελπίζω, λοιπόν, και το θέμα αυτό να σας απασχολήσει και να καταφέρετε να δραστηριοποιήσετε πιο πολύ τους Υπουργούς Υγείας για την καταπολέμηση των επικίνδυνων χημικών ουσιών. Ίσως λοιπόν θα μπορούσατε να φροντίσετε να δραστηριοποιηθούν πιο ενεργά οι Υπουργοί Υγείας προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί θεωρώ ότι πολλά θέματα προκύπτουν από τον τομέα του περιβάλλοντος, αλλά τελικά έχουν αντίκτυπο και στην ίδια μας την υγεία. Και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν οι Υπουργοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Σοφία Κονίλα, η Πρόεδρος, και μετά ο κ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί σας. Γρήγορα, γρήγορα, γιατί με συγχωρείτε καθυστέρησα, είχα μια άλλη συνάντηση που έπρεπε να παραστώ σήμερα το πρωί σχετικά με τα εφητεύματα στήθους. Να σας πω ορισμένα πράγματα, αλλά θα το κάνω ιδιαίτερα γρήγορα. Αυτό το σημείο μου φαίνεται σημαντικότατο και πρέπει να το θίξουμε. Πρόκειται για την ε, αναγνώριση και πιστοποίηση, πιστοποίηση για την εταιρεία που έθεσε αυτά τα φυτεύματα στην αγορά. Χρειάστηκε μια πιστοποίηση λοιπόν και αν κατάλαβε ότι θα ήταν στη Γαλλία πιο δύσκολη όλη η διαδικασία και πηγαίνοντας σε ένα άλλο κράτος ε, διαφορετικό θα μπορούσε να είχε μια πιστοποίηση πιο εύκολη όσον αφορά τη διαδικασία αυτή. Και σε αυτό το επίπεδο αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παρέμβουμε και μάλιστα γρήγορα γρήγορα για να πετύχουμε μια εναρμόνιση σε αυτές ε, τις διάφορες φάσεις διαδικασίας για την πιστοποίηση, ώστε παντού να ισχύουν τα ίδια σε όλα τα κράτη-μέλη σε ένα επίπεδο τέτοιο που να προστατεύει τους πολίτες και όχι τους ε, βιομηχάνους. Έτσι, αυτό ήθελα να θίξω σαν πρώτο σημείο. Ένα σημείο ακόμα σχετικά με την άθληση. Η συγγήτρια ήμουν ε, σε μια έκθεση για την άθληση και αυτό σαν μέτρο εργαλείο δημόσιας υγείας ε, και είναι κάτι που ισχύει από την εφαρμογή την 1η Δεκεμβρίου του 2009 της Συνθήκης Λισαβόνας και θεωρώ ότι τα θεσμικά μας όργανα έχουν αυτή, την, έχουν αυτή την αρμοδιότητα και για την κοινωνία και για τη δημόσια υγεία και είναι πολύ σημαντικό αυτό σε θέματα πρόληψης. Πολλά και διάφορα θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο κρατών μελών προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ, Κρατών Σένης τώρα και μετά Μισελή μαζί. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω, κυρία Υπουργέ. Σας καλωσορίζουμε σε αυτήν την Επιτροπή και προσβλέπουμε στα αποτελέσματα αυτού του εξαμήνου. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες ότι ξέρουμε πόσο έχετε προχωρήσει σε πολλά θέματα και ξέρουμε ότι μπορείτε να προχωρήσετε ακόμη περισσότερο. Θα θέσω μία ερώτηση που παρεμφερείς με αυτή τη Δάνα για τα προβλήματα τα ενδοκρινολογικά που μπορούν να εμφανιστούν. εξαιτίας αυτών των κοκτέιλ ουσιών που αναφέρθηκαν. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Δεν έχουμε τα κατάλληλα μέτρα και θα πρέπει να υπάρχει βούληση για να ληφθούν μέτρα εκ μέρους της Επιτροπής Αναφέρομαι σε διάφορα ε, προβλήματα τα οποία μπορούν να προκληθούν από ουσίες που εκλείνονται ακόμη, εκλείονται, με ακόμη και από τα έπιπλα, από τα αντικείμενα που μας ε, ε γυρίζουν, από διάφορα σκευάσματα, από τα τρόφιμα κτλ. Πέρσι είχε πει υπουργό σα ότι όλα αυτά τα θέματα θα είναι θέματα προτεραιότητας για την Προεδρία σας. Σκέπτεστε να λάβετε κάποια μέτρα, να κάνετε αναθεώρηση της οδηγίας Ρίτς ή με κάποιον άλλο τρόπο θα αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ τελευταία ομιλήτρια Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω κυρία Υπουργέ. Έχουμε μεγάλες ελπίδες και προσδοκίες. Σχέση με τις ε, αρμοδιότητες που έχετε αναλάβει και τα πρωτοβουλίες που έχετε λάβει στη χώρα σας. Πρώτη μου ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό να είστε σε συνεργαστία με τον Επίτροπο Ντάλι για τον τρόπο με τον οποίο οι διάφοροι οργανισμοί λειτουργούν. Διότι θα είμαστε αξιόπιστοι αν οι οργανισμοί που έχουμε δημιουργήσει δουλεύουν σωστά. Για τον οργανισμό φαρμάκων υπάρχει πρόβλημα σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ κάποιων κρατών και νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσει η λειτουργία αυτού του οργανισμού χωρίς να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αυτών που είναι επικεφαλής. Το δεύτερο θέμα, το μπισφενόλ. Πολλές χώρες, όπως το Βέλγιο και η Γαλλία, ίσως και η Δανία, έχουν απαγορεύσει τη χρήση του μπισφενόλ. Τι θα κάνετε σε επίπεδο Ευρώπης, και αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τη λειτουργία της ΕΦΣΑ, του οργανισμού φαρμάκων, θα πρέπει αυτό τι την ε, ουσία να την απαγορεύσουμε για όλα τα σκεύη που αν θέλετε βρίσκονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Προς το παρόν έχει απαγορευτεί τα μπιμπερό των μωρών. Αλλά πρέπει να προχωρήσετε. Τρίτη παρατήρηση. Υπάρχει με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία πρόβλημα. Όπως ξέρετε όλοι και περισσότερες αντένες υπάρχουν στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις που καταδικάζουν την προσέγγιση τους, τι θα κάνετε. Σήμερα το πρωί έχουμε ένα σεμινάριο για τα παιχνίδια που περιέχουν τοξικές χημικές ουσίες. Τι θα κάνετε. Στα πλαίσια λοιπόν της αναθεώρησης διαφόρων οδηγιών θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ώστε να γίνει υποχρεωτική η απαγόρηση χρήσης αυτών των απαράδεκτα ε, επικίνδυνων ουσιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε και τώρα περνάμε στις απαντήσεις. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή την πραγματικά ανοιχτή συζήτηση. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις διάφορες ερωτήσεις που μου τέθηκαν. Ε, κύριος Νικόλα είπατε ότι οι γυναίκες δεν είχαν κατανοήσει τον κίνδυνο των εμφυτευμάτων στήθους. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι και οι ιατροί έχουν ευθύνη απέναντι στις ε, ασθενείς πελάτησές τους. Θα πρέπει να τους εξηγήσουν ε, και δεν ξέρω γιατί ε, ε, οι πολίτες θα πρέπει να λάβουν εκείνη την ευθύνη για όσα γίνονται μετά από ιατρικές ενέργειες. Βέβαια το σημαντικό θα είναι οι ίδιες οι γυναίκες να αποφασίσουν για το τι επιθυμούν αφού πρώτα ενημερωθούν κατάλληλα για τους κινδύνους. Περιμένουμε την πρόταση της Επιτροπής προς στιγμή και γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή προωθεί μια απόφαση για να αντιμετωπίσει το θέμα των ευμητευμάτων στήθους που αποτελούν πια σκάνδαλο σχετικά με τις διάφορες διατάξεις ιατρικές και το που θα ισχύουν ε, περιμένουμε την απάντηση και έχουμε και τους διάφορους κωδικούς όλα αυτά. Ελπίζουμε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση και να συνεργαστούμε με Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Το θέμα τώρα του καπνού, του καπνίσματος. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη αυτό ακριβώς αφορούσε η ερώτησή σας. Αν θα πρέπει να ενισχύσουν την όλη νομοθεσία. Ναι, η νομοθεσία σχετικά με τον καπνό, το κάρσμα είναι σημαντική και λυπούμεθα γιατί κανείς δεν προχωράει περισσότερο όσον αφορά τα θέματα αυτά. Θα προσπαθήσουμε να το προωθήσουμε και στη Δανική Προεδρία και σχετικά Κύριε Νικόλα, για αυτό το θέμα που μιλήσατε, σίγουρα ε, διεξάγονται συζητήσεις ε, σχετικά με το ισχύει σε διάφορες χώρες ε, και μέλη της Επιτροπής σας έχουν ζητήσει να συζητηθούν αυτά τα θέματα με την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη και εμείς ακούμε τις διάφορες απόψεις έστω κι αν δεν είναι από τις προτεραιότητες που εξέφρασα πριν από λίγο. Κύριε σχετικά με την φαρμακοαντίσταση των μικροβίων, στα αντιβιωτικά δηλαδή κυρίως, ε, ναι, θα απαιτηθεί, συμφωνώ, μια ολιστική αντιμετώπιση. Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια, θα πρέπει να ανταλλάξουμε τα στοιχεία μας, τις πληροφορίες μας. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να προσέχουμε και ακόμα για... Ε, ξέρω ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Κύριε Όκεν. Ναι, μπορείτε να χαρείτε και ο γιος σας θα είναι εδώ μαζί μας ε, σε λίγο και θα ήθελα εγώ ίδια να είμαι παρούσα για τη συνάντηση στη συνάντηση αυτή. Ελπίζω ότι υποβάλλετε ερωτήματα, αλλά για το πώς επηρεάζουν τα φάρμακα την υγεία και το πώς αυτά μπαίνουν στο περιβάλλον κλπ. Σίγουρα είναι σημαντικό το θέμα. Δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιου χαρακτήρα και θα πρέπει οι Υπουργοί επίσης περιβάλλοντος να συζητήσουν μαζί μας για το πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και το παιδί σας ακριβώς είναι ο αρμόδιος υπουργός. Λοιπόν, ακούστε ε, το να είναι αποτελεσματική μια διαδικασία, όλα αυτά δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος του καταναλωτή, του ασθενούς, στα πλαίσια του καλύτερη υγεία, καλύτερη ζωή. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει, να ισχύσει αυτή η καινοτομία, να ισχύσει αυτή η ανάπτυξη. Συμφωνούμε λοιπόν με τη σφαιρική αντιμετώπιση και όσον αφορά τις χρόνιες ασθένειες. Για τον κύριο Σεν, Μπορώ να σας λέω με το όνομά σας. Νταν, έτσι. Λοιπόν, σχετικά με το συσσωρευτικό αποτέλεσμα αυτό το κοκτέιλ, όλα αυτά στο Δανικό Κοινοβούλιο τα συζητήσαμε και προσέχουμε ιδιαίτερα αυτό το συσσωρευτικό αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό και οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Υγείας να συζητήσουν από κοινού το θέμα και το πρόβλημα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και λαπιδράσεις που είναι δυνατές εδώ. Χρειάζεται να το εξετάσουμε εάν τα πράγματα θα μπορούσαμε να τα εξετάσουμε καλύτερα έτσι, με καλύτερο πιο ήρεμο τρόπο σχετικά με όλα αυτά και ε, σε λίγο θα το πει και υπουργό Περιβάλλοντος όλα αυτά στα πλαίσια του 7ου προγράμματος Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μια λεπτομερής ανάλυση, θα δούμε και τις σχετικές, ανέργειες, τις σχετικές ενέργειες με τις χρόνιες ασθένειες και το διαβήτη. Ναι, για την Κρίστελ, Κρίστελ θα μπορούσα να τα πείτε επίση αυτά. Δεν είναι άμεσα αρμοδιότητας ε, αλλά θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε το θέμα πιο έξυπνα. Προσπαθούμε να τα δούμε επίσης κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας Θεωρώ ότι θα χάναμε μια ευκαιρία ε, να γνωρίζαμε περισσότερα πράγματα για την κατάσταση και θα ήταν ανόητο από δική μας πλευράς να μην το κάνουμε λοιπόν. Κύριε Βάις Γκέρμπερ, σχετικά με την ενημέρωση των ασθενών. Ήδη το ανέφερα ότι η Προεδρία μας επιθυμεί να ξεφύγει από το σημερινό αδιέξοδο. Θα πρέπει όμως το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να ακολουθήσουν μια στάση, να υιοθετήσουν μια στάση επικοδομητική και να προσπαθήσουν και εκείνοι να βρουν μια διέξοδο. Θα το κάνουμε και εμείς από τη στιγμή που το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι έτοιμα να συνεργαστούν μαζί μας. Και για την κυρία Βέστλουν τώρα, για την ε, φαρμακοαντίσταση των μικροβίων είναι κάτι το πολύ σημαντικό, συμφωνούμε μαζί σας και θα πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Είναι από τις προτεραιότητες, να επαναλάβω, της Προεδρίας και παίζουν ρόλο ταυτόχρονα και το περιβάλλον και η υγεία κλπ. Και, και έρχομαι εδώ στο δεύτερο ερώτημά σας. Όπως είπα στον Ταν Γιώργενσεν, είναι κάτι το οποίο μελετάμε, άλλωστε συμφωνούμε με όλες αυτές τις προτεραιότητες και θα μπορούσαμε να εντατικοποιήσουμε την εργασία και στα πλαίσια ενός διαλόγου. Η κυρία Οκόνη. σχετικά με τα εμφυτεύματα στήθους. Ε, ναι, θα πρέπει να ενημερωθούμε αμοιβαία, συμφωνούμε και η Επιτροπή να την απασχολήσει ιδιαίτερα και επίσης σχετικά με την άθληση σίγουρα είναι σημαντική για τη δημόσια υγεία και κατά γενικό τρόπο θα πρέπει να βοηθήσουμε στον τομέα αυτό και με τα όσα είπατε συμφωνούμε. Τι άλλο έχουμε? Ο κύριος Αρσένης. Αυτό που είπατε, ναι. Όχι. Μπισφανόλη Αλφα όχι. Ποιος τι. Νομίζω ότι απάντησα στην κυρία Οκόνη. Ο κύριος Αρσένης, ναι, ναι, ναι, για τον κύριο Αρσένη. Όπως σας έλεγα. Ναι, το περιβάλλον και η υγεία είναι πολύ σημαντικά. Θα πρέπει να δούμε πώς αυτά τα δύο μπορούν να συνδυαστούν και όταν άκουσα το ερώτημά σας, Αναρωτήθηκα μήπως ήταν κάποιος ε, επίδεσε ερώτηση γιατί ε, το γνωρίζετε εγώ ακριβώς ε, είπα στο Δανικό Κοινοβουλίο ότι την πισφενόλη Α θα πρέπει να την απαγορεύσουμε στα μπιμπερών. Λοιπόν σε μένα προσωπικά είχατε απευθυνθεί. Πάντως και υπουργό Περιβάλλοντος θα σας επιβεβαιώσει σε λίγο ότι είναι μια τρομερά πλατιά συζήτηση σχετικά με όλο αυτό το συνδυασμό και είναι μέρος του 7ου προγράμματος, προγράμματος δράσης, κάτι το πολύ σημαντικό. Και για να τελειώσουμε τώρα, η κυρία Ριβάζη. Ζητήσατε μια συνεργασία με τον Επίτροπο, ναι. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε διάθεση να συνεργαστούμε με τους Επιτρόπους με τον Επίτροπο στην περίπτωση αυτή, αλλά θα πρέπει να διαθέτουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό πολύ σημαντικός ο διάλογος αυτός. Μίλησα για τη Βυσφενόλη Α και για τα παιχνίδια. Ίσως να αφήσω την ε, Υπουργό Περιβάλλοντος να απαντήσει γιατί νομίζω ότι από την μέρος της αρμοδιότητάς της αλλά σίγουρα χρειάζεται το περιβάλλον και η υγεία να συνδυαστούν στις προσπάθειές μας και είναι πολύ σημαντικό αυτό για τα παιδιά που είναι μια ομάδα υψηλού κινδύνου απέναντι στο πρόβλημα αυτό και σημείωσα πάντως όλες τις παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής σας και χαίρομαι ιδιαίτερα για τα σχόλια που άκουσα, τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις που μου υποβάλατε και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Χαίρομαι όμως ε, προκαταβολικά για αυτή τη συνεργασία δεν έχω καμία αμφιβολία για το επικοδομητικό πνεύμα το οποίο θα ισχύσει. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω πραγματικά για την παρουσίαση, γιατί πραγματικά είσαστε η αρμόδια υπουργό ε, Υγείας, ασκείτε χρέη Υπουργού Υγεία, αλλά και Υπουργού ε, Μπορικής Πολιτικής. Με δύο λοιπόν οι μα μας μιλήσατε και τα καταφέρατε εξαιρετικά. Μας δείξατε τι έχει πρόθεση να κάνει η ιδανική Προεδρία σε όσα μας παρουσιάσατε, με όσα μας παρουσιάσατε πρέπει να πω ότι δημιουργήσετε μία συμμαχία προθήμων εδώ, στο Κοινοβούλιο. Θέματα όπως η ενημέρωση των ασθενών που συχνά μας προκαλούν μεγαλύτερη αγανάκτηση παρά μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Θα τα βάλετε στο επίκεντρο της ε, δράσης σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας εύχομαι κάθε και σας παρακαλώ ε, να χαιρετήσετε και τους συναδέλφους τους οποίους εκπροσωπείτε και ενημερώθηκα ότι σήμερα το απόγευμα θα παρατεθεί και στην Επιτροπή Εμπορικών Υποθέσεων και η Επιτροπή αυτή ασκεί πολιτική που έχει να κάνει με το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερα για την Βανική Προεδρία. Να ξέρετε ότι είμαστε πάντα στο πλευρό σας για όλα όσα μας παρουσιάσετε. Θα υπάρχουν ασφαλώ ε, διαστάσει απόψεων σε κάποια επιμέρου στοιχεία, αλλά σε γενικέ γραμμέ θα ήθελαμε να σα πω, θα θέλαμε να σα πούμε ότι είναι άριστα προετοιμασμένη η Προεδρία σα και σα ευχόμαστε ότι καλύτερο και προσβλέπουμε στη συνεργασία μα του επόμενου έξι μήνε. Ευχαριστώ. Μάλιστα λοιπόν, να περάσουμε στο σημείο 22 της ημερήσιας διάταξης, στο 6ο Παγκόσμιο Φόρουμ για το νερό στη Μασαλία, 12 με 17, με 22, συγγνώμη, Μαρτίου, λέει ο Πρόεδρος. Και εδώ θα εγκρίνουμε μια προφορική ερώτηση θα ήθελα καταρχάς να δώσω το λόγο στο Ρίχαρτ Ζίπερ και να τον συγχαρώ γιατί έχει τη γραφειά του. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τις ευχές σας. Να σας, σας παρακαλέσω η Σοφή Οκονή, η οποία συνέταξε την, μαζί μου το ψήφισμα, να πάρει πρώτο το λόγο. Μάλιστα, πολύ ωραία η Σοφία Κονή, λέει ο Πρόεδρος στη Μασαλία στη λαμβάνει χώρα και νομίζω ότι είστε και υπεύθυνοι για θέματα Μασαλία. είναι λοιπόν πρέπει και αρμόζουν. Euh, Ευχαριστώ που μου δίνει το λόγο. Πολύ κομψή κίνηση εκ μέρου, σου, αλλά δεν με εκπλήσει. Όντω. σήμερα η ιδέα είναι να παρουσιάσουμε το ψήφισμα που σας έχει διανεμηθεί. Το σχέδιο ψηφίσματος αυτό έχει σχέση με την οργάνωση αυτού του Παγκόσμιου Εβδόμου Φόρουμ για το νερό που οργανώνεται φέτος στην Μασαλία από τις 17 έως 22 Μαρτίου. Πιστεύουμε εμείς μέλη της Επίτροπη Περιβάλλοντος, του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να υποφεληθεί από αυτό το παγκόσμιο γεγονός για να στείλει ένα σαφέστατο μήνυμα στο σύνολο των ε, πολιτικών και όσων συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα. Να στείλουμε λοιπόν ένα ισχυρό και ηχηρό μήνυμα όταν θα λάβει χώρα αυτό το φόρουμ. Γι' αυτό έχουμε την πρόταση ψηφίσματος αυτή, την οποία υποστηρίζει το σύνολο των πολιτικών ομάδων, οι σοσιαλιστές, οι πράσινοι, οι άλντε, οι γκούε. Θα αφήσω λοιπόν τον Ρίτσαρντ να σας παρουσιάσει το θέμα από την δική μας οπτική γωνία. Παρουσιάζουμε τέσσερα μεγάλα θέματα που είναι οι τέσσερις διαφορετικές, τα τέσσερα διαφορετικά κεφάλαια τα οποία θέλησαν κυρίως να προωθήσουν οι οργανωτές αυτού του φόρουμ. Πρώτα απ' όλα, ευημερία για όλους, εξασφάλιση ευημερίας για όλους, Δεύτερον, συνεισφορά στην ε, οικονομική ανάπτυξη. Ας κάνουμε μπλε τον πλανήτη μας. Και τέταρτο κεφάλαιο, ποιες είναι οι συνθήκες που πρέπει και οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να μπορέσουμε να επιτύχουμε. Θα ήθελα να περιμήσω στα πλαίσια αυτής της πρώτης ψηφίσματος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια είχαν μια πάρα πολύ καλή πολιτική σε θέματα προβληματικής για το νερό. Λαμβάνουμε υπόψη τους στόχους οι οποίοι τέθηκαν από τον ΟΗΕ που θεωρούν ότι το νερό είναι ένα κοινό αγαθό για όλη την οικουμένη. Ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Ανθρώπινο δικαίωμα για τον καθένα από εμά να έχει πρόσβαση σε πόσιμο είδωρ. 800 όμως εκατομμύρια άτομα δεν έχουν πρόσβαση σε νερό ε, πόσιμο, καθαρό, έτσι. Ή έχουν πρόσβαση δηλαδή σε ακάθαρτο νερό. Και 2,5 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας ε, της έλλειψης μη ποσίμου ύδατος. Λαμβάνοντα λοιπόν όλα αυτά τα θέματα υπόψη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στο σύνολο των ε, μετεχόντων. Εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με δική του πρωτοβουλία εδώ και 30 χρόνια οργανώνει τις χώρες οι οποίες έχουν ε, τις υδάτινες λεκάνες και Ξέρουμε ότι η πραγματογνωσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια ανταλλαγής καλών πρακτικών και συνεργασιών αποκεντρωμένα μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται ώστε όσοι ζουν πέραν των συνόρων μας να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο νερό και πιστεύω ότι πρέπει με την ε, αποκεντρωμένη συνεργασία πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε την χρηματοδότηση ε, για το νερό σε διάφορες χώρες πριν ε, Ευρωπαϊκής, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε ώστε στις χώρες μας να συνεχίσουν να υπάρχουν τα κατάλληλα προγράμματα εξυγίασης των υδατίνων πόρων που έχουν δικαίωμα να έχουν όλοι οι πολίτες μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εμένα με Απασχολείται για το θέμα αυτό. Άλλωστε έκανα και τη διπλωματική μου στο θέμα αυτό. Μπορούμε λοιπόν πάρα πολύ να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Αλλά για να πάρουν το λόγο όλοι οι συναδέλφοι θα ήθελα να περιοριστούμε όλοι σε 1,5 λεπτό γιατί οι δεν θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε μέχρι τις 11.30 που θα έρθει να μας επισκεφτεί η υπουργό. Ο Ρίχαρτ Ζέμπερ να πάρει το λόγο ως ε, συνεισηγητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και ιδιαίτερα την Σοφή που εργάστηκαν στο θέμα αυτό. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας βοήθησαν ε, στην ε, σύνταξη του θέματος αυτού. Το θέμα λοιπόν είναι πώς θα προωθήσουμε τον τομέα αυτό. Δυστυχώς η κατανάλωση νερού αυξάνεται κατά διπλάσιους ρυθμούς από ό,τι αυξάνεται ο πληθυσμός της γης. Πρόκειται για ένα αγαθό απαραίτητο για την γεωργία και για την υπόλοιπη ανάπτυξη και νομίζω ότι η Ευρώπη θα πρέπει με την νομοθεσία της να συνδράμει προς την επίλυση του προβλήματος. Μετά από αυτά που είπε η Σοφή θα ήθελα να αφήσω το χρόνο για τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα από τους Ελληνικοκράτες λέει ο Πρόεδρος, ο κ. Ζάμπο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρόβλημα του νερού είναι πρωταρχική σημασία. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν. Και είναι ένα από τα θέματα για τα οποία θα μιλήσουμε στο Παγκόσμιο Φόρουμ για το νερό. Το μήνυμα λοιπόν Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό. Θα πρέπει να διατηρήσουμε την ε, δομή αυτού του κειμένου ώστε να αποστείλουμε ένα σαφές και συνοπτικό μήνυμα. Μιλούμε για κάτι που είναι ε, πρωταρχικό, θεμελιώδες δικαίωμα παγκοσμίω για όλους και νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι ότι όντως είναι ανθρώπινο δικαίωμα και κοινό αγαθό το νερό. Το 2009 είχαμε αποφασίσει ότι θα πρέπει να επαναβεβαιώσουμε την θέση μας μέσω του ψηφίσματος αυτού. Εάν μιλούμε για πρόσβαση παγκοσμίως σε αυτό το κοινό αγαθό, θα πρέπει να πούμε με ποιες συνθήκες μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτό το αγαθό. Ίσως με τη χρησιμοποίηση κονδυλίων και επιδοτήσεων ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση σε αυτό το κοινό αγαθό σε κάποιες πάρα πολύ πτωχές περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πολύ λίγο χρόνο στη διαθεσή μου και θα επανέλθω αργότερα με άλλες παρατηρήσεις της συζήτησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Ζεμπράντη για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ μάλλον και τους συναδέλφους που ανέλαβαν την πρωτοβουλία για το, για το ψήφισμα αυτό. Είναι θετικό το ότι το Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό καθίσταται ένα παγκόσμια κλίμακα φόρουμ όπου συζητιούνται θέματα περί του νερού, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά ασφαλώ και το συνειδητοποιούμε όλοι. Θα ήθελα να τονίσω κάποια ζητήματα τα οποία θα ήθελα να προσθέσω στο ψήφισμα. Ένα είναι η σημασία του γεωργικού τομέα, γιατί αποτελεί το βασικό ε, τομέα κατανάλωσης νερού και το βασικό τομέα που μολύνεται άλλωστε και το νερό στην Ευρώπη. Μπορούμε λοιπόν να κερδίσουμε πάρα πολλά αν επικεντρωθούμε στον τομέα της γεωργίας. Ένα άλλο ζήτημα είναι το εξή. Χτες συζητήσαμε θέματα βιοπικιλίας. Είναι σαφές ότι το καθαρό νερό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για την βιοπικιλότητα, αλλά και αντίστροφα. Είναι σαφές ότι πρόκειται για τις μία από τις πιο σημαντικές υπηρεσίε που μας παρέχει η φύση. Το καθαρό νερό στην ε, Ολλανδία, για παράδειγμα, στη χώρα μου, έχουμε αμόλοφους και καθαρίζεται το νερό μέσω των αμόλοφων και ρώτησα την βιομηχανία του ύδατος, τι θα μας κοστίσει αν δεν υπήρχαν αυτοί οι αμόλοφοι και θα πρέπει εμεί να προβούμε σε καθαρισμό του νερού. Πραγματικά εκατομμύρια και εκατομμύρια. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ακριβώς αυτούς τους δύο τομείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τώρα η Σάτου Χάση για τους πράσινους. Okay, then Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σχέδιο αυτό είναι αρκετά πλήρες κατά την απόψή μου και συμπεριλαμβάνει τα διάφορα θέματα που τίθενται, θέματα που τίθενται για την διαχείριση του νερού και στο ξεκίνημα από που προέρχεται αλλά και που καταλήγει και επίσης τις διάφορες απόψεις ε, όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητά του βέβαια. Ίσως να υποβάλουμε μια προσθετική παράγραφο, μια τροπολογία στα πλαίσια αυτής της σύνταξης που είναι θετική, καλή κατά την απόψή μας. Ένα μηχανισμό ακριβώς όσον αφορά το, τις τιμές που θα ισχύουν γιατί πάει... Ε, αντίθετα από αυτό που έπρεπε. Όσο περισσότερο νερό χρησιμοποιεί κανεί, τόσο λιγότερο πληρώνει το κυβικό. Και κυρίως στη Γεωργία, στη Γαλλία είναι το 80% της κατανάλωσης νερού που γίνεται από τους γεωργούς, αλλά πληρώνουν λιγότερο αυτή την χρήση νερού και την ε, χρηματοδότησή του. Άρα λοιπόν ε, μία τροπολογία θα υποβάλουμε για μια καλύτερη, δικαιότερη επιβολή τιμών, ε, σωστό, δίκαιο για να αποφύγουμε τη σπατάλη νερού και να παροτρύνουμε τον κόσμο να μην σπαταλάει το νερό μέσω ενός κατάλληλου μηχανισμού τιμών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επόμενος Επόμενη μιλήτρια, η κυρία Γιάννα Σέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ για την εκλογή σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Σεβέρ και την κυρία Οκονή που πρότειναν την πρόταση ψηφίου τους αυτή που θεωρώ ότι είναι πλήρης στα πλαίσια του δυνατού ξεκινούμε από το κεκτημένο ότι το νερό είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα βασία. Δεύτερον, επιμένουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, δομημένα σχέδια ανα υδρολογική λεκάνη και νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε ακόμη περισσότερο ώστε να δοθεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό, όπως λέγεται το σημείο 11, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το οποίο λέμε για χρόνια. Δηλαδή ότι οι τοπικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους ένα ποσοστό του φόρου που επιβάλλεται στο νερό για να μπορέσουν να προωθήσουν συνεργασία σε περιφερειακό τοπικό επίπεδο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει στα πλαίσια αυτού του φόρου να δούμε πώς θα μπορέσουν οι διάφορες αρχές και οργανώσεις ε, που έχουν ήδη εκφράσει την βούληση για αυτό τον φόρο να συμφωνήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε αυτό το ψήφισμα πιστεύω θα μπορούσαμε να έχουμε πιο συγκεκριμένα σημεία. Ξέρουμε ότι έκανε πάρα πολλά πράγματα και καλά η Κομισιόν για το νερό. Είναι όμως κάτι διαφορετικό αυτό που γίνεται τώρα. Κάναμε δηλώσεις, δηλώσεις και τώρα πρέπει να περάσουμε στις λύσεις, τις συγκεκριμένες, γιατί ε, όλοι ξέρουμε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα με το νερό. Όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ε, ολοκληρωμένη πολιτική μεταξύ βιοπικιλότητας, γεωργίας και νερού. Μιλούμε για τις τιμές, αλλά οι τιμές εξαρτώνται από το πού προέρχεται η τιμή και πώς διοχετεύεται. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ε, αυτό που συμβαίνει στη Νότια, στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για γενική πολιτική ύδατος. Και το ε, κόστος καθαρισμού επίσης είναι διαφορετισμό. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ελέγξουμε με διαφάνεια το θέμα της προέλευσης. Γιατί εκεί βρίσκεται η μεγάλη διαφθορά όσον αφορά το νερό. Απ' την άλλη θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η νέα διαχείριση είναι κάτι στο οποίο αντιτίθενται πολλές χώρες, όπως η Τουρκία Φερρυπίν. Ώστε, διότι ξέρουμε ότι από διάφορες υδρολογικές λεκάνες και ποτάμια εξαρτώνται πολλές χώρες. Υπάρχουν κάποιες ε, ε, πολιτικές και μάχες που είναι χαμένες. Ας μην ε, ε, συνεχίζουμε χωρίς να προχωρούμε με ρεαλισμό για λύσεις. Ευχαριστώ. Ο Βιτόριο Πρόντι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σύντομα, ιδιαίτερα σύντομα, σαν μέλος της ομάδας εργασίας ε, για την προσαρμογή και την αντιμετώπιση της κλιματολογικής αλλαγής θα πρέπει να πω το θέμα το πώς θα προσέξουμε το περιβάλλον και να διατηρηθεί το νερό εκεί που συγκεντρώνεται στην αρχή όσο γίνεται περισσότερο και να μπορέσουν και τα υπόγεια να γεμίσουν σε εισαγωγικά. Και αυτό μετά και στις αστικές περιοχές η αντιμετώπιση γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αδιαβροχοποίηση που αν δεν γίνει προκαλεί ιδιαίτερες απώλειες. Εδώ να τονίσω και τη σημασία λοιπόν του εδάφους για να εξοικονομήσουμε νερό γιατί είναι ένα σύνολο το οποίο πραγματικά επιτρέπει ή όχι να έχουμε την κατάλληλη διαχείριση του νερού που να είναι σωστή και αποδεκτή. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι είναι σημαντικό το νερό και επειδή δεν έχουμε πολύ νερό και όχι μόνο στην Μασαλία αλλά και αλλού θα πρέπει να το δούμε και σε διεθνούς χώρους και συναντήσεις για να το μεταπαιδεύσουμε κατάλληλα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κουκοβιτσιά, ένα λεπτό από εδώ και πέρα. Πρόεδρε, ζητάω συγγνώμη εάν ε, μακρηγόρησε κάπως πριν από λίγο. Εγώ θα ήθελα περισσότερη προσπάθεια στο ψήφισμα αυτό να εκφράσουμε αυτή την άποψη, ώστε στην Ευρώπη να πίνουμε περισσότερο νερό από τις βρύσες μας χωρίς να είναι κίνδυνος για την υγεία μας. Ευχαριστώ. κυρία Κρίστα Κλάσε ευχαριστώ, μιας και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο δεν μπορούμε να αναφερθούμε εκτενώς σε θέματα για το νερό, αλλά νομίζω ότι σημαντικά, είναι σημαντικό να μην επανεφεύρουμε τον τροχό. Άκουσα από τους ε, βασικούς συζητητές ότι όλα αυτά που αναφέρθηκαν συμπεριλήφθησαν και στην ε, σχετική έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα που αφορούσε και θέματα για το νερό. Σω θα πρέπει να τα κοιτάξουμε εκ το κείμενο αυτό. Μάλιστα, πολύ ωραία λέει ο Πέδρος. Θα πρέπει να ψηφίσουμε ποιοι είναι υπέρ του ψηφίσματος για το νερό. Κατά. Μάλιστα, εγκρίνεται λοιπόν. Να ψηφίσουμε το σχετικό ψήφισμα στις ε, θα ψηφίσουμε 29 Φεβρουαρίου, 1η Μαρτίου εδώ στην Επιτροπή μας το ψήφισμα και στην 1η του Μαρτίου θα ψηφιστεί το ψήφισμα αυτό στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και να περάσουμε στο επόμενο θέμα και καλωσορίσουμε την Υπουργό. Να καλωσορίσουμε λοιπόν ε, την Ίντα Άουκεν, ασκούσα χρέη Υπουργού Περιβάλλοντος, ε, μάλλον ασκούσα χρέη ε, επικεφαλής του Συμβουλίου και Υπουργού Υπουργό Περιβάλλοντος της Δανίας. Είναι πραγματικά οικογενειακή συγκέντρωση σήμερα. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμά σας. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο Ακούσαμε την ε, παρουσίαση της ε, Υπουργού, πολύ καλά προετοιμασμένη. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, γιατί ανυπομονούμε να ακούσουμε την παρουσίαση εσά, να ακούσουμε την ε, πλευρά της Δανικής Προεδρίας. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο και μετά θα, ακολουθήσουμε, θα ακολουθήσει ένας γύρος ερωτήσεων, γιατί έτσι ήθιστα. Δύο γύροι ερωτήσεων συγκεκριμένα, γιατί θα είναι πολλέ οι ερωτήσει. Να ακούσουμε όμω καταρχά την παρουσίασή σα. Έχετε το λόγο. Äh, σα ευχαριστώ στα γερμανικά, Υπουργό, ε, κύριε Γκρότε, και σα εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σα. Νομίζω ότι προσβλέπω πραγματικά στην ε, συζήτησή μα και συνεργασία μας. It's Έχω την τιμή και την ευχαρίστηση να αναφερθώ σήμερα στις ε, ε, πρωτοβουλίες της Δανέζικης Προεδρίας για τους επόμενους ε, Προσβλέπουμε σε καρποφόρη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργανών. Να σας διαβεβαιώ κύριε Πρόεδρε ότι η Δανέζικη Προεδρία είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί πολύ στενά μαζί σας. Εάν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι διαφορετικό στα θέματα του περιβάλλοντος πρέπει να συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όλους τους παίκτες. Πρέπει να είναι μια κοινή προσπάθεια αυτό που θα κάνουμε. Έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες διότι γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκές οικονομίες πλήττονται από την δημοσιονομική κρίση που απειλεί όλη την Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα σημείο εκκίνησης δύσκολο για μας Προεδρία. Είμαι όμως πεπισμένη ότι η ανταπόκριση στην παρούσα κρίση δεν είναι το σενάριο business as usual δεν πλήθεται μόνο από δημοσιονομική κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπόλοιπε χώρε του κόσμου πρέπει να αντιμετωπίσουν την κρίση των πόρων και την κλιματική αλλαγή. Και όλε αυτέ οι κρίσει είναι αλληλοσυνέντετε και θα, μεταξύ του και θα πρέπει να τις επιλύσουν, επιληθούν με συνεκτικό τρόπο δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις στην οικονομική κρίση αν δεν μπορέσουμε να επιτύχουμε οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη αν δεν αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Και για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα πρέπει επίσης να βελτιώσουμε και την αποδοτικότητά μας όσον αφορά τις πηγές που χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα βελτιώσει μόνη την ανταγωνιστικότητα και τα ωφέλη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η αποτελεσματική χρήση των πόρων που διαθέτουμε και είναι ο μόνος δρόμος για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε με ε, αηφόρο τρόπο τις φυσικούς πόρους που διαθέτουμε. Και δεν μιλώ μόνο για τους ενεργειακούς πόρους, μιλώ και για την ενέργεια, για τις πρώτες ύλε, για το έδαφος, τον αέρα, την βιοπικιλότητα και το νερό. Πρέπει να μπορέσουμε για να επιτύχουμε αυτό να κάνουμε πιο πράσινη την οικονομία μας και πιστεύω ότι η πράσινη αλλαγή της οικονομίας, οικονομίας μας είναι ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε και απαραίτητος. Χρειαζόμαστε ε, μία, ένα πολιτικό πλαίσιο, ένα πολιτικό πλαίσιο που θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες τις οποίες θα μπορέσουν να αναπτυχθούν και να προχωρήσουν η καινοτομία και η αποδοτικότητα των πόρων μας. Αυτές οι οικονομικές δυνατότητες και η ασφάλεια της παροχής των πόρων μας ε, θα επιτευχθούν αν έχουμε την κατάλληλη νομοθεσία, design στα προϊόντα μας, ή κοκαινοτομίες και αηφόρο διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου που διαθέτουμε των φυσικών πηγών πλούτου που έχουμε τις δυνατότητες ανακύκλωσης, ανάκτησης και αλλαγής και αντικατάστασης κάποιων υλικών που χρησιμοποιούμε. Και αυτά είναι στοιχεία κλειδιά για την πολιτική περιβάλλοντος μας. Για την Προεδρία μας είναι μεγάλη προτεραιότητα να κάνουμε την πολιτική περιβάλλοντος ένα κεντρικό παίκτη της μετάβασης σε μια πράσινη Ευρώπη. Ε, θέλουμε να υπάρχει ε, η προσέγγιση της αποδοτικότητας των πόρων ως ένα από τα βασικά στοιχεία που θα συζητήσουμε στην διάσκεψη του Ρίο και για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και να φτιάξουμε το νέο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Το νερό, το καθαρό νερό, το πόσιμο νερό είναι ένα μεγάλο παράδειγμα. Είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε και στο διάσκεψη του Ρίου και ελπίζουμε ότι θα μας ε, θα δημοσιεύσει την μελέτη της η Κομισιό για την διασφάλιση των υδατίνων πόρων της Ευρώπης. Για μένα η διάσκεψη του Ρίο είναι είναι πραγματική ε, δυνατότητα που έχουμε ώστε να πάρουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρουμε, είναι η κινητήρια δύναμη στο θέμα αυτό και σπρώχνει τους πάντες ώστε να υπάρχει μια πιο πράσινη οικονομία βασιζόμενη στην κεντρική πρόταση του ε, έγινε στον οδικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μου κάνω ό,τι μπορώ για να βελτιωθεί η κατάσταση και να ενισχυθεί η θέση της Ευρώπης πριν από τη διάσκεψη. Η Προεδρία μας θα προετοιμάσει τις, ε, ε, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών για το Περιβάλλον του Μαρτίου θα συζητήσει τα θέματα του ε, Ρίο στην Δανία και θα ε, φτάσει στο Ρίο με συγκεκριμένα ε, προτάσεις. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να αναλάβουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις ώστε να μπορέσουμε στην, να βοηθήσουμε στο θέμα αυτό. Ε, η ατζέντα του Ρίου. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει η ατζέντα αυτή να μπορέσουμε να συζητήσουμε ε, διάφορα θέματα που είναι σημαντικά, όπως αυτό του να αφήσουμε σιγά σιγά, να εγκαταλείψουμε σιγά σιγά την χρησιμοποίηση κάποιων ε, επιδοτήσεων που είναι βλαπτικές για το περιβάλλον. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε στα πλαίσια Τη διάσκεψη του Ρίου να ασχοληθούμε με θέματα όπω η ενέργεια, το νερό, η γεωργία, η δυτική πολιτική, το θέμα των αηφόρων ανεπτυγμένων πόλεων. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν να γίνουν ε, πάρα πολύ σημαντικά ε, βήματα στη Διάσκεψη του Ρίου στην ε, περιοχή μας, όπως ξέρουμε, ε, εμείς στην Ευρώπη έχουμε ένα διαστρατηγικό στρατηγικό ρόλο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να μας βοηθήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο να παρουσιάσουμε, ε, να προπαρασκευάσουμε την θέση μας για την διάσκεψη αυτή. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να μας υποστηρίξετε. Εκτός από το Ρίο Συνήκωση, θα πρέπει να ασχοληθούμε και αυτό είναι μία από τις μεγάλες προτεραιότητές μας, με την ε, εκπόνηση του εβδόμου σχεδίου δράσης για το περιβάλλον. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας ε, ε, βοηθήσει να προχωρήσουμε και αυτό είναι ένα από τα κύρια θέματα που θα ασχοληθούμε. Χαιρετίζω επίσης το οδικό χάρτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής πίσε για την αποδοτικότητα των πόρων που θα πρέπει να αποτέσει ακρογωνία λίθος το 7ο αυτό πρόγραμμα. Η χρησιμοποίηση των ε, βελτιωμένων προϊόντων, ε, αποδοτική παραγωγή, το να κάνουμε μία ε, σωστή χρήση και προστασία του φυσικού κεφαλαίο που διαθέτουμε. ποικιλότητα, νερό, αέρας, ε, υγιή, ορυκτά προϊόντα, υδάτινη πόρη, είναι μεγάλη, είναι η μεγάλη ευκαιρία την οποία έχουμε. Πιστεύω ότι αυτό το νέο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να λειτουργήσει με τρόπο συνεκτικό ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αποδοτικότητα των πόρων. Κατά την άποψή μου, αυτό το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να εστιαστεί σε συγκεκριμένα θέματα. Τη ετήσια έκθεση της ε, Οργανισμού για το Περιβάλλον το 2010 ε, αποδεικνύει ότι δεν ξεκινάμε εκ του μηδενός, διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν ήδη στα θέματα αυτά προωθημένη ε, πολιτική και νομοθεσία. Υπάρχει λοιπόν κάτι στο οποίο να μπορούμε να βασιστούμε για να προχωρήσουμε. Εκτός από την αποδότηκα των πόρων, νομίζω ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε και νέες πολιτικές στον τομέα του κλίματος, κυρίως σε θέματα προσαρμογής κλιματικής, ε, θέματα που αφορούν την υγεία και την οδηγία REACH, όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα των ε, ενδοκρινικών διαταρακτών μεταξύ άλλων. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε γενικότερα να κάνουμε την οικονομία πιο πράσινη. Θέλουμε να πούμε ότι στην ε, ε, οδικό χάρτη της Κομισιό βρίσκουμε πάρα πολύ σωστές προτάσεις και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ώστε να μπορέσουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε θέματα κοινή αγροτικής πολιτικής και κοινή αλληλευτικής πολιτικής να βελτιώσουμε πολλά πράγματα για την ε, προστασία του περιβάλλοντος, της φύσης και την βιοπικιλότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα δημοσιονομικά ε, προγράμματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε η δική μας ε, ε, προσέγγιση θα πρέπει να είναι ρεαλιστική αλλά και φιλόδοξη. Η πράσινη ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει και η κατάλληλη υποστήριξη εκ μέρους του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αν αυτά γίνουν πραγματικότητα προς όφελος των ε, πολιτών της Ευρώπης. Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω πάρα πολύ σύντομα τους διάφορους φακέλους στους οποίους θα ασχοληθούμε προτεραιότητα κλειδί για μας είναι να μπορέσουμε να έχουμε έναν ηγετικό ρόλο αποτελεσματικό στο Συμβούλιο και για να μπορέσουμε να αναλάβουμε διαπραγματεύσει με εσά για τα διάφορου φακέλου που έχουμε επιτάπητο. Θέλουμε να προωθηθούν οι διαπραγματεύσει για του διάφορου φακέλου στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό και να φτάσουμε να καταλήξουμε σε πολιτικές συμφωνίες κατά διάρκεια της Προεδρίας μας θα συνεχίσουμε τις δραπραγματεύσεις, τέσσερις προτάσεις που κληρονομήσαμε από την, πολιτική, από την Πολωνική Προεδρία. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, για να δώσουμε την δυνατότητα στις χώρες που το επιθυμούν ή να απαγορεύσουν να μειώσουν την χρησιμοποίηση τέτοιων προϊόντων και την καλλιέργειά τους. Εξετάζουμε τη δυνατότητα ε, να ξεμπλοκάρουμε την ε, μειοψηφία που μπλοκάρει τα πράγματα στο Συμβούλιο, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε, ε, αυτό στοχεύουμε, σε πολιτική συμφωνία στο ε, Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος στο Μάρτιο. Ξέρω ότι για τα θέματα του περιβάλλοντος τα θεωρείτε ιδιαίτερα σημαντικά εσείς. Θα κάνω ό,τι περισσότερο μπορώ, ώστε να μπορέσω να βρω συμβαστικές λύσεις σε θέματα πάρα πολύ σημαντικά που αφορούν κυρίως την απαγόρευση των περιορισμών χρήσης των γενετικά τροποποιημένων ε, προϊόντων. Ελπίζω επίσης ότι θα μπορέσουμε κάτι να κάνουμε για το θέμα των, ε, της αναθεώρησης της οδηγίας που αφορά την έκκληση φύου από τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στα πλοία θα θέλαμε να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο εάν δεν μπορέσει να γίνει δυνατή πρώτη ε, συμφωνία μετά την πρώτη ανάγκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ως ελάχιστο να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το πρωτόκολλο 6 στην Σύμβαση Μαρπόλ. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν το γεγονός ότι οι εκπομπές θείου από τα πλοία το 2020 θα είναι περισσότερα από τις ε, εκπομπές ε, ε, άλλων αερίων σε χερσαίο επίπεδο και ότι 50.000 πολίτες της Ευρώπη πεθαίνουν πολύ ενωρίς κάθε χρόνο εξαιτίας της μόλυνσης από το θείο, πιστεύω ότι πρέπει για την πρόταση αυτή να είμαστε πάρα πολύ ε, φιλόδοξοι. Επίσης, αναδιατύπωση του κανονισμού ΠΙΚ που αφορά την ε- εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χημικών ουσιών. Θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε πρώτη ανάγνωση συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι αν λάβω υπόψη ε, τις ψηφοφορίες που έλαβαν χώρα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος υπάρχουν προοπτικές να καταλήξει συμφωνία. Τώρα, η οδηγία σε Βέζο 3 είναι η τελευταία πρόταση την οποία κληρονομήσαμε για τον έλεγχο πολύ σημαντικών ατυχημάτων και κινδύνων ε, εξαιτίας ε, της, ε, των επικίνδυνων αυτών ουσιών. Αρχίσαμε να δουλεύουμε για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο μόλις άρχισε η Προεδρία μας και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τις συμβαστικές λύσεις που θα μας επιτρέπουν να ξεπεράσουμε την, το πρόβλημα που δημιουργείται από την μειοψηφία που μπλοκάρει τα πράγματα στο Συμβούλιο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε συμφωνία στα πλαίσια πρώτης ανάγνωσης. Τώρα, κανονισμός, νέες προτάσεις από την Επιτροπή, κανονισμός του Δημοσιονομικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης για το LIFE, το πρόγραμμα LIFE 2014-2020. Ε, πρόκειται για την ε, πρώτη πρόταση για την περίοδο 2014-2020 που αφολείται που αφορά θέματα σε εφαρμογή του Natura 2000, είναι το πρόγραμμα Life μέλος του πολιετούς δημοσιονομικού προγράμματος και η Ιδανική Προεδρία ελπίζει ότι θα μπορέσει να προχωρήσει ε, το φάκελο αυτό. Ε, επίσης, ε, το δεύτερη, δεύτερη μας πρόταση αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στο υδάτινο περιβάλλον. Το τρίτο αφορά πρόταση για την καταστροφή παλαιών πλοίων. Ελπίζω τελικά να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σε επίπεδο Συμβουλίου σε δύο πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Το COP11 για την βιοπικιλότητα και τις ε, ε, διαπραγματεύσεις για τον ε, και το σείσμε. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε λοιπόν να προχωρήσουμε πάρα πολύ ε, τα θέματα αυτά. Λαμβάνοντας υπόψη την ε, παγκόσμια κρίση, πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ενωμένα και να μπορέσουμε να συζητήσουμε την κινητοποίηση των πόρων μεταξύ όλων και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών το οποίο θα οργανώσουμε για το θέμα αυτό ε, στο Συμβούλιο του Μαΐου. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτη σε παγκόσμιο επίπεδο η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση σε θέματα βιοπικιλότητος και θα προσπαθήσουμε ε, να προχωρήσουμε όπως μπορούμε. Επίσης ε, υπάρχει το θέμα των διαπραγματεύσεων για τον υδράργυρο και θέλουμε η επόμενη σύμβαση να είναι ε, πάρα πολύ, που είναι πόσο σημαντική, να μπορέσει να προχωρήσει, δεδομένου ότι ξέρουμε ότι ο υδράργυρος μεταφέρεται ε, από τον αέρα και το νερό και μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνος για την υγεία. Επιτρέψτε μου στα συμπεράσματα να πω συνοπτικά ότι η φιλοδοξία μας είναι να έχουμε μια αποδοτική και επαγγελματική προεδρία. Θέλουμε να δείξουμε το δρόμο για μια νέα κοινοτική πολιτική περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε μπροστά μας ε, την δυνατότητα να συνεργαστούμε στα πλαίσια μιας ανοιχτής προεδρίας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, τις, ε, έχουμε μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πράσινες τεχνολογίες και αηφόρο καινοτομία για να βοηθήσουμε την οικονομία μας. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε μεταξύ μας για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε την παγκόσμια ατζέντα. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να προωθήσω την δουλειά που μου έχει ε, που πρέπει να επιτελέσω. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποδεχθεί την προσκλήση μου να βάλουμε από κοινού τις δυνάμεις μας για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμα που μας παρουσιάζεται και είναι σαφής, ε, σαφές ότι πνέει ένας νέος άνεμος εδώ στην αίθουσα. Οι συνάδελφοι, είμαι σίγουρος, θα έχουν πάρα πολλές ερωτήσεις να σας θέσουμε. Έχουμε 14 συναδέλφους οι οποίοι ήδη έχουν ζητήσει το λόγο. Χρονικό πρόβλημα λοιπόν διαπιστώνω εκ νέου. Δύο λεπτά θα πρέπει να περιοριστούμε. Στα δύο λεπτά θα πρέπει να περιοριστούμε και θα, ε, με περιορίσω, θα κλείσω και το κατάλογο μιλητών. Να διαβάσω τα ονόματα. Kahnbach, dann der Kollege Gabrandi, dann die Kollegin Sadrine Bellier, Karl-Heinz Floren, Orsa Westlund, Vittorio Prodi, Jolanta Hibner, Karl Schlüter, Christa Klaas, Dan Jörgensen, Sofia Marcel Kukovic, Jo Lein, Kriton Asenis und Satu Hassi. Ist nicht vergessen worden. Also beginnt. Δεν σας ξεχάσαμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με το Richard Zeber. 10 λεπτά για την Προεδρία και δύο γύροι ομιλητών για ερωτήσεις. Ξεκινάμε με το, Richard, με το Richard Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ γιατί καταφέρατε να επαναφέρετε και τα θέματα ισότητας φύλου. Έχουμε εξίσου πολλές γυναίκες όσο και άνδρες στις υπουργικέ θέσεις. Είναι μεγάλη χαρά αυτή να βλέπουμε νέες ε, δυναμικές γυναίκες σε φακέλους και υποθέσεις όπως το περιβάλλον. Νομίζω ότι έχετε την απαραίτητη εμπειρία. Δεν ήξερα ότι συνδέεστε οικογενειακά και Νομίζω ότι ήσασταν σε πολύ καλά χέρια για τη συζήτηση αυτή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ε, και στη μία θα παρευρεθείτε στη συζήτηση. Η κυρία Υπουργό θα μας παρουσιάσει τα θέματα αυτά στην σχετική αίθουσα που καταφέραμε να κλείσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στα θέματα ΚΑΠ και περιφερειακής πολιτικής αναφέρατε θέματα πολλαπλής ε, συμμόρφωσης, που θέλετε να τα ενισχύσουμε αυτά σε ό,τι αφορά και την οδηγία για το νερό. Τι φαντάζεστε ότι θα γίνει συγκεκριμένα. Θα αναπτυχθούν συγκεκριμένοι δείκτες και πώς μπορεί η πολιτική μας να διαμορφωθεί με πιο φιλικό τρόπο για, για το νερό. Μία ερώτηση για τις ε, γεννητικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Θα ξέρετε ότι υπάρχουν δυσκολίες εδώ. Πώς ε, θα διαλυθεί αυτή η μειονότητα η οποία σήμερα μπλοκάρει τα πράγματα στο Συμβούλιο. Τελευταία ερώτηση για τους δεσμευτικούς στόχους σε ό,τι αφορά την ενεργειακή υποδοτικότητα. Δεν είναι ακριβώς δικό σας το θέμα, αλλά πώς δημορφώνεται η κατάσταση στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάλμπαχ και μετά η κυρία Ζεμπραντή. Ναι, θα είμαι κι εγώ σύντομη. Μιλήσατε για τη βιοπικιλότητα διαφορές. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Κατάλαβα ότι είσαστε ότι είστε υπέρ των θεμάτων για τους γενετικούς τροποποιημένους οργανισμούς. Πολύ θετικό αυτό. Η πολιτική για την βιοπικιλότητα στον γεωργικό τομέα. Πού θεωρείτε ότι υπάρχουν ευκαιρίες. Ακούσαμε τι μας είπε και η Υπουργός ε, Γεωργίας δεν είναι μόνο, μας είπατε, μια, ένας τίτλος η βιοποικιλότητα Θα πρέπει να υλοποιηθεί. Πού λοιπόν θα θέσετε τα σημεία προτεραιότητά σας. Ευχαριστώ κυρία Κάτενμπαχ και τώρα ο κύριος Γκέρμπραντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα μόνο να ευχαριστήσω την Υπουργό Άουκεν για την παρουσίασή της, αλλά θα ήθελα και να τη συγχαρώ για το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμά της για τους επόμενους έξι μήνες. Νομίζω ότι εδώ θα βρείτε τρμή υποδοχή για τα προγράμματα σας, για τη βιοπικιλία, για την πράσινη ανάπτυξη και το καθεξής. Εγώ ανησυχώ κάπως παραπάνω για το ψυγείο που θα αντιμετωπίσετε, την παγωμάρα που θα αντιμετωπίσετε από πλευρά του Συμβουλίου. Κοιτώντα το τι κάνει, τι κάνει το Συμβούλιο για το περιβάλλον, για να είμαι διπλωματικός, πρέπει να πω ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται ιδιαίτερα θετικά. Το Δεκέμβριο το, Υπουργείο, ε, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος παρατήθηκε μπροστά στο Συμβούλιο Γεωργίας. Η αποδοτικότητα των πόρων δεν έχει ακόμα σφαγιαστεί στο Συμβούλιο, αλλά η θερμή υποδοχή των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει πραγματοποιηθεί πραγματικά. Ο νέος λοιπόν φρέσκος αυτός άνεμος που πνέει στη Δανία, πώς θα μεταφραστεί ανησυχώ όταν θα μπει στους κόλπους του παγωμένου Συμβουλίου. Και σε καιρούς όπου είναι τόσο σαφές ότι χρειάζονται βιωσιμότητα για την οικονομία μας, όχι μόνο επειδή μοιαζόμαστε για τον πλανήτη σας. Τι θα γίνει. Τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαντρίν Μπελιέ και ο Καλχάιτς Φλόρεντς. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ. Και εγώ, όπως και οι συναδελφοί μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας δώσω συγχαρτήρια για το τόσο φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα. Δύο-τρεις τομείς ε, θα με απασχολήσουν ε, για μερικές διευκρινήσεις. Είπατε από τις προτεραιότητές σας ε, τη σύμβαση στη Δανία πριν από 10 χρόνια, Δαρούς, ε, για την ενημέρωση του κοινού και τη συμμετοχή του και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Από το 2003, τρίτος πυλώνας, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη έχει παγώσει στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Περιμένουμε τώρα όσο ποτέ μια οδηγία εναρμόνισης για την πρόσβαση αυτή, για το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε η Δανική Προεδρία τι προβλέπει για να ξεπαγώσει η όλη διαδικασία για αυτή την οδηγία, τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να ενεργήσουν, να δράσουν για το δίκαιο όσον αφορά το περιβάλλον να μπορεί να ισχύσει πριν από το τέλος του 2012 και εμείς οι οικολόγοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το υποστηρίζουμε αυτό. Επίσης αναφέρατε στο Ρίο τον Ιούνιο που μας έρχεται την συνάντηση για τον πλανήτη μας. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι περισσότερο, να μας διευκρινίσετε, να μας διαβεβαιώσετε ότι θα προωθήσετε όλα αυτά και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την συνάντηση. Επίσης θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε εάν ε, θα υποστηρίξετε στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων αυτό τη σύσταση ενός νέου παγκόσμιου οργανισμού περιβάλλοντος ε, απέναντι που θα ενταχθεί στον Παγκόσμιο, Οργανισμό Εμπορίου και επίσης θα υποστηρίξετε μια πράσινη οικονομία στα πλαίσια μιας οικολογικής αντιμετώπισης και κοινωνικής δικαιοσύνης, μια νέα οικονομία δηλαδή ο Καλ Χάιντ και μετά η κυρία Βέσλοντ. Σας ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ για τη δροσερή σας ομιλία. Είχα την τιμή να ασχοληθώ και σε κάποιες ε, ε, διαδικασίε συναλλαγή με το Συμβούλιο. Πρέπει να πω ότι η οικογένειά σα μου εμπνέει εμπιστοσύνη, αλλά αυτό σημαίνει και κάποιε υποχρεώσει. Μιλήσατε για τα θέματα γενετικώ τροποποιημένων οργανισμών ε, στα κράτη-μέλη και ότι θα πρέπει να προωθηθούν. Η συνάδελφο από την ε, Αυστρία συμφωνεί. Εγώ, κοιτάξτε, ε, έχω την ατυχία να μένω 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ολλανδία. Και διάφορε ζωοτροφέ λοιπόν εισάγονται από την Ολλανδία στη Γερμανία. Πώς λοιπόν ως μικρός εκτροφέας θα πρέπει να διαπιστώσω αν έχει γενετικώς οργανισμού ε, ιζωτροφή ή όχι. Η απόφαση είναι αυτή που είναι γιατί δεν υπάρχει πλειοψηφία. Αλλά πώς να βρει ο Γεωργός και ο εκτροφέας τι γίνεται και να μας πει ότι σας εγγυώμαι ότι δεν περιλαμβάνονται γάματα ομικρών. Δεύτερο στοιχείο που με ενδιαφέρει από 1η Ιουνίου θα πρέπει να ορίσουμε τους στόχους μας για τη μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ποιους στόχους θα επιδιώξετε, τους στόχους 20-20-20 ή θα ακολουθήσετε τη νέα μελέτη αντικτύπου για την τάση επικράτησης υψηλότερων ποσοστών στο Συμβούλιο, το οποίο και αυτό συζητιέται και είναι αρκετά αμφιλεγόμενο. Επίσης, για την αποδοτικότητα των πόρων. Πού είναι η προτεραιότητά σας. Το αναφέρατε πολύ σύντομα, συναδέλφα. Ευχαριστώ. Η κυρία Βέσλοντ. Και μετά Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μας παρουσιάζετε μια τέτοια μοντέρνα εικόνα για την Ευρώπη ως ε, υπουργό της Δανίας και οι γονείς σας άλλωστε έχουν συμβάλει τα μάλλα στην ε, πολιτική την ευρωπαϊκή και νομίζω ότι πολλοί θα κερδίσουν αν μιμηθούν τον τρόπο εργασίας σας. Ε, χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ, χάρηκα που άκουσατε και την παρουσίασή σας. Μας αναφέρετε πολλά στοιχεία στο πρόγραμμά σας, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά και για εμάς. Ασφαλώς, εξετάσαμε το πρόγραμμά σας ε, για την Προεδρία και ε, σε ό,τι αφορά τις επιδράσεις των κοκτέιλ, σε ό,τι αφορά τα θέματα νανοηλικών νομίζω ότι αποτελούν θέματα τα οποία έχει επεξεργαστεί εκτεταμένα η Δανία και νομίζω ότι θα πρέπει να απασχολήσουν και τις επόμενες γενιές. Θα πρέπει λοιπόν να δραστηριοποιηθούμε και ασφαλώς και θα σας υποστηρίξει και το Κοινοβούλιο. Ελπίζω να σας υποστηρίξουν και οι άλλοι υπουργοί προκειμένου να προκύψουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα Βικτωριο Πρόντι η κυρία Χίμπνερ και μετά θα ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος ερωτήσεων και θα ακούσουμε την Υπουργό. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Υπουργό γιατί η παρουσίαση της περιέλαβε πολλά, πάρα πολλά θέματα. Να ρωτήσω κάτι. Εάν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί μια αναθεώρηση της οδηγίας ε, για το περίβλημα, για αυτές τις σακούλες, τις πλαστικές ε, που ε, εξαφανίζονται από μόνες τους. Γιατί τι γίνεται, θα υπάρχουν και άλλες οδηγίες για τους ε, άλλες σακούλες ε, που διατηρούνται επί μακρόν στο περιβάλλον και ακόμα μπορούμε να υπολογίζουμε στη Δανία για να ξεπαγώσει αυτή η οδηγία στο Συμβούλιο τόσο σημαντική για τις ε, βιοαποδομήσιμες σακούλες και θα θέλαμε επίσης να υποστηριχτούν να υποστηρίξουμε ορισμένα πράγματα που θεωρώ σημαντικά. Πρώτα απ' όλα τις περιορισμένες φυσικές πηγές που είναι περιορισμένες. Θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα πράγματα για τη χρήση αυτών για να έχουμε μια αποτελεσματικότητά τους και επίσης όσον αφορά την αναγνώριση ενός ανθρώπινου δικαιώματος για ίση πρόσβαση στις φυσικές πηγές. Και ακόμα κάτι, για να ζητήσουμε στα πλαίσια της συνάντησης του Ρίο αυτό το κοινό αγαθό, τον ορισμό του, αυτός ο ορισμός αποτελεί την βάση για να αλλάξουν τα πράγματα στην κοινωνία μας για μια πραγματική αηφορανάπτυξη. Δύο λεπτά ακριβώς. Η κυρία Χίμπνερ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό. Είναι πραγματικά ιδιαίτερα φιλόδοξο το σχέδιο το οποίο μας παρουσιάσατε. Ελπίζουμε ότι στο τέλος του εξαμήνου θα έχετε ακόμα περισσότερους φίλους, ε, και θα πρέπει βέβαια να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε προβλήματα. Αναγνωρίσατε την αξία, τη σημασία των καινοτομιών στα πλαίσια της χρήσης των πόρων. Έτσι θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα τις πηγές αυτές και να αποτελεί και ένα κινητήρα μια κινητήρια δύναμη κατά της κρίσης. Θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε ποιες είναι αυτές οι καινοτομίες, ε, παραδείγματος χάρη και στην περίπτωση του νερού, στη διαχείρισή του, που θα μπορούσε το νερό να είναι ένα ενεργειακό στοιχείο και με μια αύξηση της μη παραδοσιακής χρήσης νερού. Και κάτι ακόμα, μια ερώτηση. Όταν μας λέτε ότι θα, πρέπει να υπάρξουν αυτές οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οι επικίνδυνες για το περιβάλλον. Τι αφορούν αυτά τον τομέα της ενέργειας ή και άλλους τομείς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Υπουργό για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Thank you very much, Uh, first uh, Ευχαριστώ συνάδελφε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Ζέμπερ, να ευχαριστήσω και τον κύριο Φλόρεντς που έφτασε τους οικογενειακούς δεσμούς. Νομίζω ότι θα περιοριστώ στα οικογενειακά εδώ. Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή και σας ευχαριστώ που μιλήσατε για την ομάδα που θα συζητήσει το θέμα αυτό σήμερα το απόγευμα. Με ρωτήσατε για την ΚΑΠ. Πώς μπορούμε να βρούμε τα χρήματα οικονομικά μέσα τα οποία θα χρειαστούν για την ΚΑΠ σε ό,τι αφορά την Ατούρα και για την οδηγία πλαίσια. Πολύ σύνθετο ερώτημα. Γιατί Κάθε χώρα αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις σε ό,τι αφορά την προστασία των ε, περιοχών Natura, αλλά ασφαλώς θα θέλαμε να υπάρχει όσο πιο πολύ πράσινος χαρακτήρας γίνεται. Αλλά και σε ό,τι αφορά το 7% ε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η φύση προστατεύεται καλύτερα σε μεγάλε εκτάσει. Δεν θέλουμε 7% εδώ και εκεί. Θα πρέπει να βρούμε και πιο ευέλικτου μηχανισμού. Και αυτό θα μπορούσε να ισχύει και για την βιοπικιλία, γιατί κάποιο έθεσε το ερώτημα. Επίση, θέσατε σημαντικές ερωτήσεις για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και πώς θα μπορούσαμε να άρουμε αυτή τη μειοψηφία που μας μπλοκάρει. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο και βλέπουμε παραπάνω από 20 χώρες που έχουν την δυνατότητα να πούν όχι στους γάματάφα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να συνεχίσουμε να το παλεύουμε. Έχουμε σε αυτή τη στιγμή μία πρόταση για τα διεκτόνα. Θα πρέπει να εξετάσουμε κατά περίπτωση κάθε προϊόν για να δούμε κατά πόσον η χώρα θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον εκάστοτε ετούντα για να εξαιρέσει την ε, εκάστοτε χώρα από την αίτησή του. Αν απαντήσει αρνητικά ο ετούντα, θα πρέπει να υπάρχει μία διαδικασία. Κατά δεύτερον, κανείς δεν θέλει να υποτιμήσει και να υπονομεύσει την έφυσα στο θέμα αυτό. Η αρχή της έφυσα δεν υπονομεύεται, κανείς δεν το επιθυμεί αυτό. και ό,τι χρησιμοποιείται για απαγόρευση γάματα φόμικρον θα πρέπει να γίνεται συμπληρωματικά προς την ΕΦΣΑ. Γιατί είναι δύσκολο να αντιταχθούμε ο ένας τον άλλον σε θέματα υγείας. Μπορεί να έχουμε συγκεκριμένα συμφέροντα βιοπικιλίας, περιβάλλοντος, αλλά αν θα μπορούσαμε να θέσουμε συγκεκριμένα τα επιχειρήματα για κάθε κράτος μέλος, αυτό ενδεχομένως να μπορέσει να άρει τη μειοψηφία. Αλλά ε, θα είναι δύσκολη διαδικασία, αλλά είναι πάνω από 20 χώρες αυτές που θέλουν να επιβληθεί η απαγόρευση. Και αυτό αποτελεί λοιπόν σημαντικό επιχείρημα. Θα δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε. Επίσης θέσατε ένα θέμα ενέργειας. Θα πρέπει να πω ότι αυτό είναι θέμα για τον συνάδελφό μου, για τον Μάρτιν Κιντεγκάρτ που ήταν εδώ χτε. Μου θέσατε το ερώτημα για την βιοπικιλία. Νομίζω ότι προσπάθησα να απαντήσω για το πώ θα πρέπει να βρούμε χρηματοδότηση στο εσωτερικό τη ΚΑΠ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ψάξουμε και άλλες πηγές χρηματοδότηση. Μαζί με τον Επίτροπο καλέσαμε τους ε, υπουργούς για την εναλλακτική εξέβρεση πόρων για την προετοιμασία για την ΚΑΠ σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ενδεχομένως και οι μελλοντικές προεδρίας να πρέπει να αναζητήσουν καινοτόμους μηχανισμούς ε, χρηματοδότησης της βιοπικιλότητας στην Ευρώπη, γιατί δεν έχουμε ακόμη α, καταλήξει. Όταν μιλήσαμε για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, Είδα την έκθεσή σα Πού είναι ο κύριο Γιώργο Λάινεν. Είδα την έκθεσή σα κύριε Λάινεν. Νομίζω ότι συμφωνήσαμε επί των βασικών θεμάτων στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Θα πρέπει να, να δούμε και τους στόχους για την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα, την προσαρμογή, τη βιοπικιλότητα και το περιβάλλον. Να δούμε λοιπόν πώς αυτά μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου. Σίγουρα θα μας απασχολήσει αυτό επισταμένος. Ο κύριος Γκερμπραντή. Πού είστε, σας βρήκα. Σας ευχαριστώ που αναγνωρίζετε ότι πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ζεστή και θερμή η υποδοχή και ξέρω ότι μας αναμένουν κρυαντούς στο μέλλον. Αυτή είναι η δουλειά μας όμως ως πολιτική. Να πιστεύουμε σε αυτά που λέμε και να συνεχίσουμε τον αγώνα. Και να συνεχίσουμε να ζητούμε επιχειρήματα τα οποία δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς. Στον τομέα λοιπόν αυτό για την πράσινη ανάπτυξη θεωρούμε ότι υπάρχουν τεράστιες ε, ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις ακόμη όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους πόρους, αλλά και για το νερό. Ξέρουμε ότι θα επενδυθούν 3 εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια στις υποδομές υδροδότησης σε όλο τον κόσμο. Το ίδιο ισχύει και για την ενέργεια. Αυτό λοιπόν είναι ένας προφανής λόγος για το ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στον τομέα αυτό. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα πριν από κάποιες οι μέρε ε, προειδοποίησαν ότι δεν θα πρέπει να περικοπούν οι, οι προπολογισμοί σε όλους τους τομείς και ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι επενδύσει στην ανάπτυξη. Και ο πράσινο τομέα είναι πραγματικά ένας τομέα όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη. Γιατί υπάρχει μεγάλο δυναμικό ανάπτυξη τη αγορά. Υπάρχουν δύο κρίσεις ε, και ίσως η περιβαλλοντική κρίση να είναι ακόμα πιο σημαντική, γιατί αν δεν την επιλύσουμε θα συνεχίσει να επανέρχεται. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσω να δώσω μια δροσερή νέα πνοή στο Συμβούλιο. Η κυρία Μπηγέ για τη συνθήκη του Όρχους. Και εδώ έχω κάποιες σχετικές υποχρεώσεις που με βαρύνουν ιδιαίτερα, αλλά ξέρω ότι προσέχετε κι εσείς ε, την ε, συνθήκη του όρχους. Θα πρέπει να σας πω ότι για την οδηγία αυτή ξέρουμε ότι είναι τεράστια η μειονότητα που μπλοκάρει το θέμα αυτό στο Συμβούλιο, αν είναι καν μειονότητα. Άρα θα πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες στην Προεδρία μας και να πούμε ότι κοιτάξτε δεν θα είναι μια οδηγία αυτή στην οποία και θα, θα επικεντρωθούμε, γιατί θεωρούμε ότι θα σπάσουμε τα μούτρα μας. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό ότι δεν θεωρούμε ότι η οδηγία αυτή δεν είναι τόσο σημαντική. Ότι δεν είναι στην ατζέντα της Δανίας αυτής, αυτή η προτεραιότητα. Απλά πρέπει να θέσουμε κάποιες προτεραιότητες. κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει ένα WEO. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Φυσικά το υποστηρίζουμε, αλλά δεν ξέρουμε αν θα υποστηριχθεί ευρέως. Θα το θέσουμε όμως στις προτεραιότητές μας, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σημαντικό θεσμικό όργανο σε θέματα περιβάλλοντος. Μπορείτε λοιπόν να μας εμπιστευτείτε. Θα δούμε τι υποστήριξη θα λάβει το θέμα για την υποστήριξη της πράσινης οικονομίας. Νομίζω ότι αυτό καταλάβατε ότι θα το υποστηρίξουμε. Δεν χρειάζεται να κάνω να επαναληφθώ. Ο κύριος Φλόρεντς έφτασε το ερώτημα των γάμα ταφ ομικρών και το σημαντικό ερώτημα του τι να κάνει ένας Γερμανός ε, καλλιεργητής εκτροφέας αν ε, χρησιμοποιούν οι Ολλανδοί από δίπλα του γάμα ταφ ομικρών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα αυτό και θα πρέπει να συνεχίσουμε να το συζητάμε. Δεν πρόκειται να επιληθεί εύκολα, δεν θα επιληθεί καν σε ό,τι αφορά αν επιληθεί αυτή η μειοψηφία. Να έχετε υπόψη λοιπόν ότι δεν έχει επιληθεί το θέμα αυτό, αλλά θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε αυτά που αναφέρει η οδηγία και η πρόταση της Επιτροπής ε, για τους στόχους 2020 είναι θέμα του Υπουργού Ενέργειας. Νομίζω ότι εκτενώς αναφέρθηκε σε αυτά χτες. Τα θέματα ενεργειακή αποδοτικότητας, σημεία επικέντρωσης. Αν θέλουμε να δούμε την Ευρώπη συνήκωση, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάποιους τομείς. Θα πρέπει να βρούμε, θεωρώ, σαφείς ε, στόχους ε, για το νερό και την ενέργεια. θα πρέπει να θέσουμε ε, και στόχους για την πατάλη νερού μέσα των συστημάτων, γιατί είναι αρκετά σημαντικός ο όγκος που χάνεται. Θα πρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία για να διασφαλίσουμε τους υδάτινους πόρους. Και είναι σημαντικό να δούμε κατά πόσον το 7 πρόγραμμα πλαίσιο μπορεί να είναι συγκεκριμένο για θέματα πόρων θα βοηθούσε πολύ να υπάρχει κάτι παρόμοιο με την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό. Να υπήρχε λοιπόν κάτι παρόμοιο και ίσως προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να εργαστούμε για να δούμε τι, ποσοστή, τι στόχοι μπορούν να τεθούν και τι ποσοστό στόχων έχουν επιτευχθεί σε τελική ανάλυση. Γιατί τώρα, για παράδειγμα, χάνουμε όλες τις σπάνιες γέες, για παράδειγμα. Ξέρουμε ότι η Κίνα κατέχει το 95% και ξέρουμε ότι είναι αδύνατον προς το παρόν να αφαιρέσουμε αυτές τις σπάνιες γέες από τα προϊόντα όταν χρησιμοποιηθούν. Πώς μπορούμε λοιπόν να σχεδιάσουμε προϊόντα προκειμένου να μπορούμε να αφαιρούμε στη συνέχεια τα απαραίτητα στοιχεία. Κυρία Βέσλουν, σας ευχαριστώ και εσάς για τη θερμή υποδοχή σε ό,τι αφορά τους ενδοκρινικούς διδαράκτες. Εξετάζουμε ενδεχόμενη θεώρηση του REACH, το εξετάσαμε μάλλον και καταλήξαμε, ότι, καταλήξαμε στο ότι ίσως είναι δύσκολη η χρονική συγκυρία λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω της τεράστιας πίεσης. Σας υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο φιλόδοξοι γίνεται. Αλλά θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η χρονική στιγμή για αναθεώρηση του REACH, αλλά ασφαλώς είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πάσα στιγμή να το συζητάμε. Μιλήσατε για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό στον θέμα των ε, διταρακτών αυτό. Κύριε Πρόντι, να σας ευχαριστήσω και εσάς για την οδηγία για τα απορρίμματα. Δεν έχουμε δει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακόμα. Θα δώσουμε προτεραιότητα στην ε, πρόταση αυτή όταν θα τη λάβουμε, αν φυσικά τη λάβουμε στη διάρκεια της Προεδρίας μας. Και η υποστήριξη της Προεδρίας για θέματα α, της οδηγίας ε, για το έδαφος. Την ίδια απάντηση θα σας δώσω όπως και για τη συνθήκη του όρχους, γιατί προφανώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κινηθούμε προς τα εμπρός αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, άρα θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για να μην είναι υπερβολικά παγωμένη η υποδοχή. Δεν νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι στην ατζέντα μας λοιπόν επί του παρόντος τα σχόλια για το Real Plus 20 και η μετατόπιση για τα υλικά. Διάβασα μία ομιλία η οποία εκφωνήθηκε πριν από 40 χρόνια και νομίζω ότι ήταν εντυπωσιακό. Θα μπορούσε αυτή η ομιλία να είναι σημερινή. Αν αφαιρούσαμε κάποια ιστορικά περιστατικά, θα μπορούσε να έχει εκφωνηθεί σήμερα η ομιλία αυτή. Έχουμε προχωρήσει λοιπόν πολύ σε κάποιους τομείς, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω σε ό,τι αφορά την θεώρηση των ε, περιβαλλοντικών πόρων ως κοινό αγαθό. Θα πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για το τι σημαίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι σημαίνει ποιότητα ζωής και σε ό,τι αφορά τους πόρους. Η συζήτηση είναι πιο σημαντική παραποτέ. Ο πολιτικός διάλογος λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικός και θα πρέπει να δώσουμε μια ορμή καινούρια, μια καινούρια ενέργεια στην όλη αυτή τη συζήτηση. Η κυρία Φίμπνερ. Πού είστε. Δεν θα είμαι και πιο δημοφιλής ε, υπουργό όταν τελειώσω το, την εκτέλεση των καθηκόντων μου στο Συμβούλιο, αλλά θα προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε ε, διάφορες απόψεις με, ειλικρινό, με ειλικρινή τρόπο προκειμένου να καταλήξουμε σε όσο πιο πολλούς συμβιβασμού γίνεται και να είστε βέβαιοι ότι θα το πράξουμε αυτό με τον πλέον πράσινο τον τρόπο, αλλά φυσικά πάντα έχουμε τους πρακτικούς περιορισμούς για την κοινοτομία. Με, ζητήσα, ρωτήσατε συγκεκριμένα τι είδους καινοτομία έχω υπόψη μου για τους υδάτινους πόρους. Θα το συζητήσουμε αυτό σήμερα. Νομίζω ότι και στο κάθε αυτό θα μπορούσατε να αντιδραματίσετε σημαντικό ρόλο. Ξέρω ότι σας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Θα πρέπει να εξετάσουμε τι δυνατότητες έχουμε, πώς προωθούμε τις επιχειρήσεις και τις ε, παροτρύνουμε να αναπτύξουν και τεχνολογίες προκειμένου να υπάρξει κοινοτομία. Στην Δανία έχουμε μακρά παράδοση υψηλών προτύπων στον τομέα του νερού και έχουμε κάπως πιο, πολύ ισχυρού παράγοντες σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τη διαχείριση, τον καθαρισμό του ύδατος. Θα πρέπει λοιπόν ε, το επόμενο θέμα να είναι η προσαρμογή, αν θέλετε. Νομίζω ότι αυτά λίγο πολύ καλύπτουν τις ερωτήσεις που μου ετέθησαν. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Κανένα συνάδελφο δεν ξεχάσατε. Ήταν τέλεια η απάντηση. Και να περάσουμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Με καλό Σλέτερ. Κρίστα κλάσματα. Two minutes. Okay. Yeah, thank you. Ναι, jag pratar svenska istället. Yeah. Ja. Um, jag vill ta upp hormonstörande ämnen som redan varit uppe. Du sa att du ville agera där. Ευχαριστώ. Θα επανέλθω σε κάτι που είπατε προηγουμένως. Είπατε ότι θέλετε να μιλήσουμε για νέα αξιολόγηση και η αναθεώρηση του ΡΙΤΣ είναι πολύ γενικόλογη. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ασχοληθείτε με θέματα που αφορούν τη συσσόρυψη των επικίνδυνων ουσιών και πολλά άλλα θέματα για τα οποία οι διάφορες επιχειρήσεις αποκρύπτουν τις πηγές τους και δεν ξέρουμε πώς έχει πραγματική κατάσταση. Υπάρχουν παρόλα αυτά ε, διάφοροι τρόποι για να τις αναγκάσουμε. Υπάρχουν τα πρόστιμα. Πολλά πράγματα λοιπόν επί χάρτου είναι τέλεια, αλλά στην ε, πράξη δεν είναι πάντα καλά τα πράγματα. Είπατε για κάποιο κείμενο που υπάρχει εδώ και 40 χρόνια. Πριν όμως από αιώνες κάποιος επίσης είπε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολλά χρήματα και έχουν ε, ε, ένα επίπεδο ζωής για τους οποίους δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε. Υπάρχουν όμως άνθρωποι και χώρες που είναι πιο φτωχές και χρειάζεται κάτι να κάνουμε ώστε να γίνουν τα συστήματα πιο δίκαια. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι πολύ ωραίες, έχουν πολύ ωραία τοπία, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις καταστάσεις και όλες τις καταστάσεις για να μπορέσουμε ε, να προχωρήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπία την οποία θα πρέπει να επιτύχουμε. Ευχαριστώ η κυρία Κλάς. Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ. Συγχαρητήρια μας προτείνατε ε, εδώ πάρα πολλές καλές ιδέες. Είστε νέα, έχετε ενθουσιασμό και πολύ ωραία σας ακούμε και ακούμε με πόσο ενθουσιασμό θίγετε όλα τα θέματα. Εμείς συζητούμε ε, εδώ και χρόνια για αυτά τα θέματα. Ο Γιάννη ο Σλίτερ είναι συνάδελφοι τους οποίους άκουσα και ξέρουμε ότι η Δανία είναι μια χώρα που ανέκαθεν ήταν πρωτοπόρος σε θέματα περιβάλλοντος. Θα ήθελα παρά το γεγονός ότι τα ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι, να επιμείνω στο ότι η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει μια συνεκτική πολιτική, να είμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο. Όχι διότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, να οπισθοδρομήσουμε οι περισσότεροι και κάποιοι μοναχικοί καρβαλάριδες μόνο να προχωρήσουν. Μιλήσατε για το ρίτσι, είπατε ότι δεν θέλει κανείς να ξανανοίξει την αθέρωση οδηγίες για τα εντομοκτώνα, για τα φυτοκτώνα που είναι πολλές φορές επικίνδυνα. Πώς θέλετε να ενισχυθεί η θέση της Ευρώπης και να βελτιωθεί για όλα των πολιτών μας εάν υπάρχουν ακόμη ε, ενδιασμοί και δεν θέλουν όλοι να προχωρήσουν από κοινού. Όλα τα θεσμικά όργανα και κυρίως τα αρμόδια θα πρέπει να μπορούν να προχωρήσουν. Μιλήσατε επίσης για τις ορμόνες που επηρεάζουν τη ζωή μας. Είστε διατεθειμένοι να λάβετε υπόψη σας και άλλα θέματα που μπορούν ε, φερειπίν να ε, βλάψουν την ποιότητα του ύδατος. Ακόμη και το αντισυλληπτικό χάπι που καταλήγει στο νερό είναι επιβλαβές. Τι μπορείτε να κάνετε για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για τις απαντήσεις που δώσατε και αυτά που είπατε. Δύο σχόλια. Θέλω να κάνω και μια ερώτηση μετά. Το πρώτο μου σχόλιο σε σχέση με αυτά τα οποία είπε η συνάδελφος προηγουμένω για το σωρευτικό ε, αποτέλεσμα το κοκτέιλ αυτό το περί των διαφόρων ε, ουσιών και ε, τις ε, ενδοκρινολογικούς διαταράκτες. Είπαν κάποιοι ότι δεν έχουμε τις τα απαραίτητα στοιχεία τα επιστημονικά για να προχωρήσουμε. Ίσως το να ασκήσουμε πίεση όμως στην Κομισιόν για να συλλέξει όλα αυτά τα στοιχεία είναι και αυτό κάτι που μπορείτε να το κάνετε. Τώρα, όσον αφορά το ΠΙΚ, θέμα για το οποίο εγώ είμαι υπεύθυνο και εγώ και οι σκιώδεις ηγητές προσπαθούν να προχωρήσουμε βρίσκοντας συμβαστικές λύσεις. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά τεχνικά θέματα, δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε στις διάφορες εταιρείες να στέλνουν στο εξωτερικό τις επικίνδυνες που έχουν διότι δεν κάνουν τίποτα στην Ευρώπη. Ούτε και αυτό είναι λύση. Επίσης, το θέμα του πρασινίσματος της ΚΑΠ. Το αναφέρετε το θέμα. Χθες ε, έθεσα εγώ το θέμα στην συνάδελφό σας στη ΜΕΤΕ, αλλά θα ήθελα να μου πείτε πάρα πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις εξέφραζαν την ανησυχία τους που τη συμμερίζομαι, ότι ε, θα προσπαθήσουμε αλλά θα είναι πολύ ανοιχτόχρωμα το πράσινο της γεωργίας και όχι πραγματικό πράσινο. Ποιες είναι οι αρχές που θα χρησιμοποιήσετε για να εξασφαλίσετε το ότι θα είμαστε πραγματικά βέβαιοι ότι θα υπάρξει σε θέμα προστασίας του περιβάλλοντος μια πραγματική προστιθέμενη αξία σε αυτό το οποίο θα κάνετε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να χαιρετήσω τη νέα Υπουργό, να την να συγχαρώ για το πρόγραμμά της και είμαι σίγουρη ότι σήμερα η μητέρα της είναι πάρα πολύ περήφανη για την παρουσίαση που έκανε. Η Δανία είναι μία από τις χώρες ε, φάρους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Γι' αυτό η χώρα αυτή μπορεί να αποτελέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός πραγματικό φάρο, πραγματικό παράδειγμα. Θα ήθελα να μου πείτε εάν προβλέπετε ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, γιατί μπορείτε να μας μάθετε πάρα πολλά. Επίσης, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε νέες θέσεις απασχόλησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να δείτε πώς θα μπορέσετε να δημιουργήσετε σχέσεις με τις ε, χώρες BRIC. Επίσης, όσον αφορά το eco-design, πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια ευρύτερη νομοθεσία, διότι οι παρούσες διατάξεις δεν είναι δεσμευτικές. Προβλέπονται μόνο σε ε, θελούσια βάση. Επίσης, θα ήθελα να μου πείτε, θα λάβετε μέτρα ώστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούμε να πίνουμε νερό από τη βρύση και όχι αναγκαστικά μόνον από τα μπουκάλια. Γιολάνη και μετά κύριε Σκρίτον σε ευχαριστώ αγαπητή Ίντα ή μάλιστα καλύτερα αγαπητή Υπουργέ. Σας εύχομαι και εγώ ότι καλύτερα και σας συγχαίρω για το εξαιρετικό πρόγραμμά σας. Νομίζω ότι μπορούμε να επενέσουμε την οικογένεια Άουκεν για την δέσμευσή της σε περιβαλλοντικά θέματα και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνεί όλη η Επιτροπή και νομίζω ότι αυτό θα φανεί και στην φάση της... Ε, ελπίζουμε αυτό να φανεί και στις ψηφοφορίες για το πρόγραμμα αυτό. Για το 7 πρόγραμμα πλαίσιο. Η προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μάλλον κακή. Καθυστέρησε την επεξεργασία του προγράμματος αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι χρειάζεται πολύ input και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να διαμορφωθεί ένα καλό πρόγραμμα για την βιώσιμότητα, την βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει <coughs> να αποτελέσει και μια, ένα, ένα σύνολο με την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Όπως είπατε, το... πρόκειται για ένα πρόγραμμα ε, ομπρέλα όλων των στρατηγικών, είτε πρόκειται για μεταρρύθμιση της πολιτικής ε, αλληλείας, της ε, ΚΑΠ, ενεργειακή αποθετικότητα, βιοπικιλότητα, όλα αυτά θα πρέπει να καταφέρουμε να τα διατυπώσουμε με συγκεκριμένο τρόπο στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Όπως είπατε, να επικεντρωθούμε στις ενέργειες, όχι μόνο στην παραγωγή εγγράφων στόχοι για το 2020 και ασφαλώς να αναπτυχθεί και ένα όραμα για το 2050. Όλα αυτά θα πρέπει να αναπτυχθούν με συγκεκριμένο τρόπο. Ελπίζω να προωθήσουμε και σε διαφορετικά ελλείμματα που αντιμετωπίσουμε και για να μείνουμε και στο χρονοδιάγραμμα. Μίλησε ο κύριος Γκερμπράντι για το παγωμένο ψυγείο του Συμβουλίου θα ήθελα να σας αναφερθώ και σε ζητήματα πάγου για, το, για την Ευρωπαϊκή Σύνοδο, γιατί με θέματα τέτοια θα ασχοληθούν όχι οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, αλλά οι αρχηγοί κρατών. Ίσως θα μπορούσατε να αναφερθείτε και σε αυτό. Μάλιστα, ευχαριστούμε Γιολάνη, ο Νασένης και μετά η Χάση. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να σας ευχαριστήσω και πρέπει να σας πω ότι στην Επιτροπή μας χαιρόμαστε που βλέπουμε ένα νέο άτομο πολύ ικανό σε αυτή τη θέση. Με νέες ιδέες που δεν επαναλαμβάνει αυτά που είπαν προηγούμενοι. Τρομερό λοιπόν αυτό. Και σας συγχαίρω για τις απαντήσεις που δώσατε μέχρι τώρα. Θα ήθελα να μιλήσω για το Ρίο Συνήκωση. Το Ρίο Συνήκωση είναι κατά κάποιο τρόπο ε, ένας άσος κατά τη διάρκεια σας, κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας. Είναι, είναι η δυνατότητα που έχετε να λάμψετε, να μας δείξετε τι μπορείτε να κάνετε. Και νομίζω ότι μπορούμε εάν ε, θέλουμε να κάτι το καλό, να θέσουμε τις βάσεις για να προχωρήσουμε μετά περισσότερο από όπου θα προχωρήσει ή μέχρι εκεί που θα φτάσει το Ρίο συνήκωση. 20. Ας πούμε ότι στο πρώτο σχέδιο προτάσεων έχουμε κάποια θέματα. Έχουμε μια πρώτη συνάντηση που λάβει η χώρα στη Νέα Υόρκη και ελπίζω θα εμπλουτιστεί αυτό το σχέδιο με νέες προτάσεις. Και οι προτάσεις θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν και αλλού. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, πληροφορίες τις οποίες έχω και νομίζω ότι θα μπορέσω να σας τις αποστείλω για να μπορέσετε να τις μεταφέρετε στους συμβούλους σας και να προχωρήσετε. Η κυρία Σάτου Χάση. Κυρία Υπουργέ, με μεγάλη ευχαρίστηση ακούσαμε τις δηλώσεις σας μέχρι τώρα. Χαίρομαι επίσης διότι αναφέρετε την οδηγία για το θείο στα καύσιμα των πλοίων. Υπάρχουν πολλά θέματα επιτάπητος στο Συμβούλιο που έχουν σχέμα με την κλιματική πολιτική και με άλλα θέματα που άπτονται της περιβαλλοντικής πολιτικής. Ένα από αυτά είναι τα βιοκαύσιμα και τα κριτήρια αηφορίας για τα βιοκαύσιμα. Όπως ξέρετε υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες όσον αφορά την ε, ισορροπία σε θέματα μονοξιδίου, δεδομένου ότι η παραγωγή των, για την παραγωγή των βιοκαυσίμων, αλλά και θέματα που μας απασχολούν όσον αφορά τις επιπτώσεις της βιοπικιλότητας με την παραγωγή βιομάσης και βιοκαυσίμων. Η Δανική Προεδρία έχει αναλάβει δεσμεύσεις ώστε να εργαστεί με τρόπο που θα επιτύχει αυτά τα κριτήρια αηφορίας για την παραγωγή των βιοκαυσίμων, ώστε να ξέρουμε ότι η παραγωγή τους δεν θα βλάψει το έδαφος, την βιοπικιλότητα και το περιβάλλον γενικότερα. Ευχαριστώ, Γιάννος Άλλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Υπουργέ, στην εισαγωγή σας αναφερθήκατε ότι είναι σημαντικό να τροποποιηθούν αυτές οι τρεις οδηγίες και ότι θα πρέπει να υπολογιστούν όλα αυτά. Θέλετε να πετύχουμε ε, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Αυτό αποτέλεσε στόχο και της Πολωνικής Προεδρίας. Υποστηρίζονται εδώ στο Κοινοβούλιο όλα αυτά, αλλά βλέπουμε ότι στο Συμβούλιο τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Να σας συστήσω λοιπόν. Να σας πω ότι στις διαπραγματεύσεις ε, προέκυψε το ότι δεν θα πρέπει να μειωθεί το επίπεδο ασφάλεια σε σχέση με τις σημερινές, ε, τα σημερινά ισχύουσα, ισχύοντα. Θα πρέπει λοιπόν ο τομέας εφαρμογής να περιοριστεί. Θα πρέπει να εξαιρεθούν κάποιοι τομείς. Αυτό θα μπορούσε να παρεμποδίσει μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Θα ήθελα να σας πω ότι οι συγητές και οι εμπειρογνώμονες, οι σκιώδες και εγώ ο συγητής κάνουμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να επιλύσουμε τα αμφιλεγόμενα στοιχεία, αλλά είναι πραγματικά ευαίσθητη η ισορροπία που πετύχαμε εδώ στο, Κοινοβούλιο και θα πρέπει πραγματικά να προσέξουμε από πλευρά Συμβουλίου. Ευχαριστά και προστάθηκα και εγώ ως τελευταίος στην λίστα των ομιλητών. Για το πακέτο για το κλίμα. Μιλήσαμε για τη βιομάζα και για την ε, βιώσιμη παραγωγή της. Πρόκειται για μια ελάχιστη συμβιβαστική πρόταση, κοιτώντας ότι στα κράτη-μέλη υπάρχει μια, ένας ανταγωνισμός για τις εκτάσεις. Η συνάδελφό σας για τις γεωργικές εκτάσεις, το ξέρει αυτό. Τις... Θα πρέπει να οριστεί με πιο ακριβή τρόπο το πώς παράγεται η βιομάζα με βιώσιμο τρόπο και σε θέματα ε, όταν συζητήσαμε την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, τα συζητήσαμε αυτά. Υπήρξε και μια σχετική πρωτοβουλία, ίσως θα υπάρξει μια πρωτοβουλία από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να αυξηθεί και η αποδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα βιομάζας. Προκειμένου λοιπόν να γίνει αυτό θα πρέπει να οριστούν ε, αυστηρά κριτήρια και θα πρέπει και μεταξύ των διαφόρων τομέων να μειωθεί κάπως αυτός ο ανταγωνισμός που υπάρχει γιατί στο βιοαέριο ανταγωνιστικός κλάδος είναι ο γαλακτοκομικός, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των εκτάσεων. Αν θα υπήρχε λοιπόν σχετική πρωτοβουλία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πιο αυστηρή διατύπωση των κριτηρίων αυτών, κατά πόσον θα μπορούσατε να το υποστηρίξετε αυτό στο Συμβούλιο για να ξέρουμε και εμείς που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Μάλιστα. Και έτσι ολοκληρώσαμε λοιπόν και το δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα στον κύριο Σούντερ για τους διαταράκτες. Μιλήσατε για κάποιους τομείς στους οποίους κάτι μπορούμε να κάνουμε. Και συχνά λέει κανείς δεν είδα τίποτα, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Αλλά εμείς νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε στρατηγική να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Και βεβαίως, αν είναι, είναι θέμα κονδυλίων, πάντα υπάρχει το θέμα της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε για τα θέματα αυτά είναι πραγματικά σε πρώτη φάση να βρούμε τις πληροφορίες. Να δούμε για τα σχημικές ουσίες, αφού τις εξετάσουμε και έχουμε την απαραίτητη επιστημονική γνώση, να προωθήσουμε τα πράγματα. Να δούμε Πώς μπορούμε σε κάθε χώρα να απαγορεύσουμε τη χρήση τους και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε ευρωπαϊκή απαγόρευση και να αποκομίσουμε τις απαραίτητες γνώσεις και στοιχεία από κάθε χώρα ώστε να προχωρήσει σε απαγόρευση τους γενικευμένη και η Επιτροπή. Εσείς ως Κοινοβούλιο και εμείς ως κράτη αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φέρουμε στο φως τις απαραίτητες πληροφορίες Πιστεύω λοιπόν ότι σωστά το θες το θέμα και σας ευχαριστώ. για αυτά τα οποία άκουσα ε, στα σουηδικά από τη συναδελφό σας. Ως πιστεύω ότι το θέμα της ε, σπάνης κάποιων πόρων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και οι σπάνεις κάποιων ε, από αυτές ε, τις, ε, αυτούς τους πόρους είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε πολύ σύντομα όλοι μας. Δεν είμαι νέα και θεροβάμων όταν μιλάω για αυτά τα θέματα. Είμαι πολύ ρεαλίστρια και ξέρω ότι πάρα πολλά εκατομμύρια άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα της έλλειψης σχεδόν βασικών πόρων. Θα πρέπει λοιπόν, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεδομένου ότι θα αφορά εκατομμύρια, είναι από δισεκατομμύρια ακόμα, θα πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε να διασφαλίσουμε την ε, επάρκεια πόρων ακόμη και για τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό με πιστεύω στα κάποια πράγματα και είμαι πάρα πολύ ενεργητική παρά το γεγονός ότι πολλές φορές κάποιες συζητήσεις μου φαίνονται δύσκολες. Επίσης, τον... Κάστε, θέλω να πω ότι συμφωνώ μαζί σας ότι πρόκειται για πρόγραμμα για όλη τη ζωή, αλλά πρέπει να το καταλάβει κανείς το εφόρου ζωής πρόγραμμα και να δει πώς θα μπορέσει να αλλάξει διάφορα κομμάτια αυτού. Εμείς ως Προεδρία και εσείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταλάβετε ότι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι η μετάβαση σε οτιδήποτε είναι πράσινο. Θα πρέπει να πιστέψετε ότι είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Ότι θα έχουμε μια κατάσταση η οποία θα είναι επωφελής και επικερδής για όλους. Ότι δεν απαγορεύουμε για να απαγορεύσουμε. Απαγορεύουμε για να δώσουμε την δυνατότητα να λυθούν πάρα πολλά, ε, πάρα πολλά προβλήματα μια και έξω. Πολλές ιδέες δυνατότητες λοιπόν δίδονται και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κάτι ε, κατανοήσετε. Ακόμη και αν χρειαστεί να αφιερώσουμε όλοι μας τη ζωή μας κάποιοι για να αλλάξουν τα πράγματα. Επίσης είπατε κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Να ενεργεί με μία φωνή η Ευρώπη. Να είναι δεμένη. Ακόμη και τώρα που είναι δύσκολα τα πράγματα είναι ακόμη πιο σημαντικό το να είμαστε όλοι ενωμένοι στην Ευρώπη. Είπαμε λοιπόν ότι για εμείς ε, στην Προεδρία μας θα πρέπει και να δίδουμε τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για θέματα περιβαλλοντικά, αλλά να είμαστε και ρεαλιστές, να ξέρουμε τι μπορεί να επιτευχθεί σε επίπεδο Συμβουλίου, ώστε να μην υπάρχουν ε, αποκλήσεις απόψεων τόσο μεγάλες. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα δύο στοιχεία να μπορέσουμε να τα συγκεράσουμε. Είναι δύσκολο αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να το επιτύχουμε. Ο κύριος Γιώργιος το είπε. Επίσης είπε ότι όντω για να μπορέσουμε να πείσουμε κάποιους να αλλάξουν τα πράγματα θα πρέπει εμείς να φέρουμε στο φως όλες τις επιστημονικές γνώσεις και τα στοιχεία που έχουμε για να μπορέσουν ε, να πείσουμε και την Κομισιόν να αλλάξει. Όσον αφορά τον κανονισμό ΠΙΚ, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το κατορθώσουμε αυτό και με συνεργασία να φτάσουμε σε συμφωνία. Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε πρασίνισμα. Και θέλουμε να συνεισφέρουν και οι δύο πυλώνες και με τα κατάλληλα μέσα και με την κατάλληλη χρηματοδότηση. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σίγουροι ότι θα ευρεθούν οι απαραίτητοι πόλοι και πιστεύουμε ότι θα πρέπει με ευέλικτο τρόπο να συνδυάσουμε τις δράσεις που θα αναλάβουμε και στα πλαίσια των δύο πυλώνων. Αυτά είναι κάποια από τα πράγματα τα οποία θα ήθελα να προχωρήσουμε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιτές, ρεαλιστές και τα πράσινα να τα λέμε πράσινα, αλλά όταν είναι ψευτοπράσινα να το αποκαλύπτουμε. Κυρία Κούκουβιτς. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Η ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Δεν ξέρω ε, πώς θα το βάλουμε στο πρόγραμμα. Θα το προωθήσω όμως για την... Ε, νερό που είναι το σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι είναι σωστή η πρότασή σας και έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι ένας θετικός τρόπος να, επιδείξουμε, να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι μπορούν να πράγματα να γίνουν καλά με την ανταλλαγή βέλτιστων ε, πρακτικών είναι κάτι το θετικό. Και αν έχετε ιδέες επί αυτού του θέματος, προωθήστε τις σε μένα. Θέλω να τις ακούσω. Eco-design οικολογικός σχεδιασμός. Ε, πρέπει να υπάρξει κανονισμός που να μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή. Αλλά ακόμη δεν, ε, δεν ξέρω τόσα πολλά από τεχνικής πλευράς. Και δεν μπορώ να σας πω, εφόσον δεν το ξέρω το θέμα, πώς πρέπει να το χειριστούμε, αλλά Κάποιος άλλος συνάδελφο θα το κάνει. Τώρα, θέλουμε όντως στη Δανία να προστατεύσουμε το πόσιμο είδο. Το νερό που μας δίνει πλούσιο η γη και πρέπει να το προστατεύσουμε. Εμείς έχουμε πολύ καλό λοιπόν φυσικό νερό, καθαρό νερό, πόσιμο και το εκτιμούμε. Και πολλέ άλλες χώρες το κάνουν. Θα πρέπει όμως όντως Εάν είναι καλό το νερό να πίνουμε τον κόσμο να πίνει νερό από τη βρύση και όχι να αγοράζει εμφιαλωμένο. Αλλά δεν ξέρω πώς σας πω να το επιτύχετε αυτό. Κύριε Λάινεν, όντως είναι το έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον δύσκολο. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση και εμείς και εσείς στην Επιτροπή να το προχωρήσει. Και είναι σημαντικό το ότι μπορώ εγώ να πω και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο ότι όντω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει αυτό το 7 πρόγραμμα να είναι φιλόδοξο και ε, σημαντικό για όλους. Σε ευχαριστώ λοιπόν και συνεχίστε την πίεση προς τους άλλους. Εμείς θα προσπαθήσουμε τον Ιούνιο για το θέμα αυτό να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Έχουμε χρόνο λοιπόν να προχωρήσουμε, να δείξουμε τις γενικές κατευθύνσεις και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα στον Ιούνιο. Και κάτι πολύ σημαντικό. Είπατε ότι... I think, of course, Θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη της οικονομίας με πρασίνισμα, πώς θα μιλήσουν οι Υπουργοί Οικονομικών και για το όριο 20 συν. Και όλα αυτά τα θέματα, πώς θα μπορέσετε και εσείς από τη μεριά σας να τα προωθήσετε. Θα δω, επίσης θα κάνω εγώ στο Συμβούλιο και θέλουμε όλα τα θέματα που μας απασχολούν τα συζητούν και οι Υπουργοί Οικονομικών γιατί και αυτή είναι πολύ σημαντική για τις ε, πολιτικές μας. Κύριε Αρσένη, σωστά λέω το όνομά σας, φαντάζομαι. Σας ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια και διότι τονίσατε ότι είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα θέματα που αφορούν το θα ξέρουμε περισσότερα συγκεκριμένα πράγματα σε μερικές μέρες. Το Ρίο είπατε κάποια συγκεκριμένα θέματα τα οποία θέλετε να προωθούν. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν βασιζόμενοι σε όλα αυτά τα συγκεκριμένα θέματα ε, να δούμε τι θα κάνουμε και τα θέματα τα οποία μας αναφέρατε μας ενδιαφέρουν και στείλτε μας τις πληροφορίες που έχετε. Κυρία Χάρση, σε θέματα θείου στα καύσιμα των πλοίων. Σας ευχαριστώ για το σχολείο σας. Κριτήρια για τα βιοκαύσιμα τώρα. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι θέμα δικής μου προτεραιότητας, αλλά ως Υπουργή Περιβάλλοντος θα πρέπει να πούμε στους αρμόδιους υπουργούς να προσπαθήσουν να είναι συνεκτικοί στις πολιτικές που κάνουν. Δηλαδή να μην λύνουν ένα πρόβλημα και να δημιουργούν τρία λύνοντας ένα. Αυτό αφορά την βιομάσα και τα βιοκαύσιμα. Ή άλλα ε, σχετικά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ζωοτροφές ή θέματα εσοδιάς, δασών, αναδάσεις, όλα αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και θα πρέπει από κοινού να βρούμε τρόπους για να λύσουμε τα προβλήματα που δημιουργούν. Και όντως και εγώ για αυτά τα θέματα θα ασκήσω πίεση στους συναδέλφους. Κύριος Άντερ. Μιλήσατε για το Σεβέζο 3. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο είπατε. Δηλαδή το ότι η σημερινή δέσμευση είναι πραγματική δέσμευση και συνένεση. Και βεβαίως δεν θέλουμε να υπάρχει λιγότερη προστασία για τους πολίτες της Ευρώπης. Στα πλαίσια του Σεβέζο 3 θα προσπαθήσουμε να μην κάνουμε κάτι το οποίο θα μειώσει τα επίπεδα προστασίας των πολιτών. Πρόκειται για ένα τεχνικού περιεχομένου φάκελο, αλλά κάνατε μια πολιτική φύση παρατήρηση πολύ σημαντική που τη λαμβάνω υπόψη. Νομίζω ότι κάλυψα όλες τις ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ. Αγαπητή ήταν Άουκεν, ήταν Πραγματικά τέλειες οι απαντήσεις σας. Μας ε, δώσατε όλες τις απαντήσεις που συζητήσαμε. Το μόνο που έχω να διαπιστώσω είναι ότι λάμπουν τα μάτια σας και πραγματικά έχετε όρεξη. Και ελπίζω αυτή η όρεξη να είναι κολλητική για τους ε, άλλους 26 συναδέλφους στο Συμβούλιο, προκειμένου με τον ε, φρέσκο, δροσερό αυτό αέρα να φροντίσουν για μια αλλαγή του κλίματος, γιατί είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η οικονομική, η χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση του χρέους θα επιληθεί με μια καμπή. Μια καμπή προς μια καινούργια οικονομία, μια βιώσιμη οικονομία. Εμείς ε, έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις επί της ατζέντα γιατί ζητείτε βιώσιμη αλία, βιώσιμη γεωργία και το ξέρω επειδή στην προηγούμενη ζωή μου εργάστηκα στον τομέα αυτό, ξέρω ότι με τη βιώσιμη οικονομία μπορούμε να βγάλουμε και χρήματα, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στην δική μου περιφέρεια. Προέκυψαν 15.000 θέσεις εργασίας καινούριε στον τομέα των ανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί να μην συμβεί αυτό και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα. Ήταν χαρά μεγάλη να σας υποδεχτούμε αυτή την εβδομάδα και εσάς και τους συναδέλφους σας και όπως είπα και στους ε, συναδέλφους ε, του τομέα της υγείας έχετε μπροστά σας ε, συμμάχους, πρόθυμους συμμάχους Σας εύχομαι εκ βάθους καρδίας κάθε επιτυχία για τους επόμενους μήνες και πέρα από αυτό και το όνομα Auken είναι συνώνυμο της ποιότητας. Σας εύχομαι το καλύτερο.